Καλημέρα σε όλους σας. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συνάντησή μας στην Επιτροπή Ανάπτυξη σήμερα το πρωί με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εκεί υπάρχει μια αλλαγή. Την έχει ζητήσει ο κύριος Γκέρενς για να βληθεί για τις 18 Δεκεμβρίου το σημείο 14 της ημερήσιας μας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με την Concord για στρατηγική, για τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη και να μπορέσει να μιλήσει για το θέμα αυτό στους συντονιστές το πρωί 18 Δεκεμβρίου πριν από τη συνάντηση της δικής μας Επιτροπής και αργότερα το πρωί να συζητήσει με την Κονκόρντ για τη στρατηγική ακριβώς της Επιτροπής μας ε, για τη συνοχή της πολιτικής ανάπτυξης από τη στιγμή που θα έχει εκφραστεί η υποστήριξη των συντονιστών. Ο κύριος Γκέρενς, ε, να υπενθυμίσω ότι είναι ο νέος εισηγητής μας για τη συνοχή της στρατηγικής ανάπτυξης. Ε, μήπως υπάρχει κάποιο σχόλιο, σας παρακαλώ, για το σχέδιο μερίσιας διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με το σημείο αυτό. Όχι, κανείς. Υιοθετείται λοιπόν η μερίσια διάταξη με την αλλαγή αυτή. Μισό λεπτό, ο κύριος Γκέρενς. Κύριε, κύριε έχετε το λόγο, ναι. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον ομιλητή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δέβα προσπαθούσε να πω στους συναδέλφους ότι ε, στις 18 μόλις έχουμε επιστρέψει από το Στρασβούργο και θα έχει και χιόνια μάλλον και την τελευταία φορά που ήρθαμε από το Στρασβούργο όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ήταν κλειστά, ήταν ε, τρομερές οι κλιματικές συνθήκες. Εγώ χρειάστηκα μια ολοκληρή μέρα να φτάσω στο Λονδίνο. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα να ψηφίσουμε στις 18. Και νομίζω ότι και οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ το ίδιο πιστεύουν. I think, am I right? I completely agree with Mr. Deva. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ντέβα. Monsieur Goerens, vous savez la parole να έχετε το λόγο πάλι. Α, εσείς, ναι. Ο κ. Ε, γιατί ε, μίλησε για την ε, αναβολή του 18 για να του 14 για να πάει στις 18, αλλά δεν θα διεξαχθεί ψηφοφόρια. Δεν ξέρω, δεν σας άκουσα καλά. Δεν δεν κατάλαβα καλά. Εδώ ε, χθε ε, και μάλιστα χωρίς πρόβλημα είχα πει για την Κοπενχάγη στην Κονκόρντο που υπήρχαν και βουλευτές Δανείοι για να μιλήσουμε για τη συνοχή της πολιτικής και σήμερα το πρωί ήρθα εδώ και δεν μπορούσα να είμαι δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί το πρωί με τους συντονιστές ε, γιατί είχαμε τη στιγμή που έχουμε σχεδιάσει να το εντάξουμε στη μεσιά διάταξη. Εντάξει, υπεύθυνο είμαι και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη για την αναβολή για τι 18, αλλά αυτό που δεν κατανόησε καλά κύριε Ντέβα, εσείς ε, γιατί, ποια, ποια αναβολή μιλήσατε ακριβώς. Ναι, θα το συζητήσουμε το σημείο 14 της 18 Δεκεμβρίου χωρίς όμως ψηφοφορία. Έτσι κανονικά δεν θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Τα πρακτικά τα έχετε για τη συνεδρία στις 8 και 9 Οκτωβρίου. Αν δεν ε, κάνετε κάποιο σχόλιο πριν από το τέλος της συνεδρίας θα εγκριθεί. Θα εγκριθούν τα πρακτικά. Έχουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι η ανακοινώσει της Προέδρου σας. Λοιπόν, χθε επέστρεψα από την Καμπούλ. Για την Καμπούλ Μπανκ ε, έχετε ακριβώς στο blog μου μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι από το μεγαλύτερα σκάνδαλα τα τραπεζικά με 800 εκατομμύρια ευρώ τα οποία χάθηκαν καθοδόν και δείχνει τις ευθύνες η έκθεσή μας ε, και πώς ε, ξεπλύνεται αυτό το χρήμα με το ρευστό αυτό χρήμα από την αεροπορική εταιρεία που ανήκει ακριβώς στους μετόχους ε, αυτής της τράπεζας και μέσω του δίσκου φαγητού μεταφέρθηκε τα, μεταφέρθηκαν τα χρήματα. Καινούρια μέθοδος ξεπλήματος. Ε, ναι, θα έχουμε και δεύτερη έκθεση ακριβώς με τα ονόματα ακριβώς. Έτσι. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για να δείξουμε ότι κάτι προσπαθεί να κάνει το Αφγανιστόν κατά της διαφθοράς, τη μάχη αυτή που δίνουμε, γιατί η διαφθορά είναι τεράστια εκεί κάτω. Λοιπόν, πήγαμε και στις φυλακές ε, και συναντήσαμε κρατούμενους, ε, οι οποίοι δεν είναι και οι πρώτοι παράγοντες. Ε. Δυστυχώς δεν σέβονται τις κανόνες της προσωρινής κράτησης στη χώρα αυτή. Έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες άτομα τα οποία δικαιολόγητα κρατούνται. Στον πρόεδρο Καρσάη αποστήλαμε, αφού συντάξαμε μια επιστολή, και έχουμε βάσιμες ελπίδες ε, ότι όσοι κρατούνται παράνομα στην Καμπούλ τουλάχιστον πριν από τα Χριστούγεννα θα ελευθερωθούν. Θα σας ενημερώσω δε στην επόμενή μας συνεδρίαση. Το κύριο θέμα που συζητείτε είναι η οργάνωση των εκλογών του 2014. Στις 16.000 που ψηφιζόταν όχι 16 εκατομμύρια, συγγνώμη, εκλογής με 12 εκατομμύρια γεγραμμένους ε, τρομερή, τρομερή απάτη. Γι' αυτό θα πρέπει να αργωθούν καλά οι επόμενες εκλογές και δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η οργάνωση. Πάντως και γι' αυτό θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές, τι θα κάνουμε. Αυτό το ε, όχι το ηλεκτρονικό σύστημα, μήπως το κανονικό, το συνηθισμένο, αλλά πρέπει να βιαστούμε γιατί το 2014 ίσως, ίσως δεν θα έχουμε καθόλου ψηφοδέλτια και θα πρέπει να ματαιωθούν οι εκλογές, κάτι που οπωσδήποτε θα πρέπει να αποφύγουμε. Πέρμαν. Ναι, θα το γνωρίζετε ότι ήμουν επικεφαλής των παρατηρητών για τις εκλογές του 2009. Όλα αυτά που λέτε είναι ακριβή, αληθεύουν. Τρομερές απάτες. Το 1 τέταρτο ή ήταν τρίτο των ψήφων στο πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Και δεν νομίζω ότι σεβάστηκαν πολλές από τις συστάσεις μας. πολύ δουλειά θα πρέπει να γίνει και ιδιαίτερα με ενδιαφέρει να ακούσω, να ενημερωθώ καλύτερα για τα συμπεράσματά σας. Ναι. Συστάσεις ακριβώς, ε, γιατί ανήκω ακριβώς σε ένα όργανο που έχει τη δυνατότητα να έχει benchmarks και συστάσεις να υποβάλει και μετά από αυτές τις παρατηρήσεις του 2009-2010 για να επηρεάσουμε την διεξαγωγή των εκλογών με το εκλογικό σύστημα του 2014. Θα δείτε και λεπτομέρειες στο blog μου για την αποστολή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θα ήθελε να κάνει μια κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτά. Καμία ερώτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε ένα αίτημα από τους ε, διερμηνείς, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το άλλο μικρόφωνο, γιατί κάνει παράσιτα. Nous allons passer au vote. Να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία, επομένως ε, να κάνουμε ένα τεστ με τις κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι χειρότερο το μικρόφωνο αυτό. Να το ελέγξουμε έτσι. Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τις ηλεκτρονικέ σα κάρτε. κάρτες. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορία, Ψήφισαν 24. Πολύ καλά. Alors... Για να δούμε. Συγγνώμη κυρία Ζολή που επιμένω, αλλά δεν μπορείτε να συνεχίσετε με αυτό το μικρόφωνο. Κάνει πάρα πολλά παράσιτα για τους διερμηνείς. Είναι σαν να το έχουν φάει αρουραίοι αυτό το καλώδιο.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 Λοιπόν, να ψηφίσουμε την έκθεση Κατρίν Γκρέσ ε, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονική.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 κατά απόχες εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 7 Λοιπόν, ψηφίζουμε συμβαστική 1, το δεύτερο το μέρος αυτό. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία συγκρίνεται με 6 ψήφους ε, περισσότερους το υπέρ. Τροπολογία 7, το πρώτο μέρος. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Καταπίπτει η τροπολογία 7, άρα λοιπόν δεν την ψηφίζουμε. 8. Όχι, ούτε 8. Η 10 παρακαλώ. 10 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαέξι σε δύο μέρη ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. προφορική τροπολογία. Ποια είναι χωρίς αριθμό. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τι έχουμε τώρα, τη 19, υπέρ, κατά, Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 19, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αποσύρεται 20, συμβαστική 3 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αποσύρεται 27, συμβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Δύο όχι περισσότερα. Τροπολογία 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 2 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 τροπολογία υπέρ μισό λεπτό μισό λεπτό Όχι, όχι, δεν ψηφίζουμε αυτή, αλλά την 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει. Το δεύτερο μέρος λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο μέρος 34 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Δύο περισσότερα τα όχι. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Δεύτερο μέρος λοιπόν, ψηφίζουμε. Πέρας, εγκρίνεται. 39 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για να δούμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση και μάλιστα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται.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 Συμβαστική 1 σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά Μήπως... Τι γίνεται, ακριβώς επαναλαμβάνουμε το ίδιο. σε 10 λεπτά δεν θα αλλάξουμε τις επιλογές μας. Έτσι, θα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ναι, εγκρίνεται. Τι. Ε, νομίζω ότι θα σεβαστούν όλοι οι συνάδελφοι, τους έχω εμπιστοσύνη την απόφαση αυτή. Το ίδιο είναι. Συνεχίζουμε. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, και εγώ το υποστηρίζω. Νομίζω ότι πρόκειται για ιδέα σοφή. Εγώ όμως αποφασίζω ότι θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 12 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, η 17 υπέρ, κατά, τις αποχές σας, εγκρίνεται, 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεκαεννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τρία Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 τροπολογία όχι, όχι, 24, 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29. 30. 30. Όχι. 32. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 σε δύο μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος 34. Ψηφίζουμε. Ένας μας λείπει. Κάποιος δεν ψήφισε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, ευτυχώς που έλεγξα. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 39 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Μετά από αυτές τις αλλαγές ψηφίζουμε αυτή την γνωμοδότηση. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. στιγμή. Ναι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Alors, nous allons voter... Euh, λοιπόν, ψηφίζουμε το σχέδιο ε, γνωμοδότησης, τη κυρίας ε, Σατζεντίνη για την συμφωνία και εταιρικής σχέσεις μεταξύ των κρατών Ανατολικής και Μεσημερινής Αφρικής και Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ε, πρόεδρε, διαφωνεί με την προφορική τροπολογία το ΕΛΚ. Α, μάλιστα, άρα δεν θα γίνει αυτό. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την πρώτη τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Le Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Nous votons maintenant le rapport de Madame. Τώρα ψηφίζουμε την έκθεση της κυρίας Γκρέζ για την βιοπειρατεία. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία της Επιτροπής Τζούρι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λοιπόν, ε, στο ίντα 6, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τζούρι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αν δεν το ελέγξουμε. Επαλήθευση με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τζούρι 7. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι τα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 6 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 42 αποσύρεται. Ήθελα να αποσύρω την τροπολογία, Πρόεδρε, ακριβώς. Τροπολογία 4 υπέρ. Συγγνώμη, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Χωριστή ψηφοφορία για την παράγραφο 17. Ψήφι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές Α, υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία 8. Τζούρι 1, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, και εδώ υπάρχει ένσταση. Τροπολογία 49, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. χωριστή ψηφοφορία παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Είναι τα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 10 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τζούρι 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 16 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα θα περάσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Voilà. Le vote est clos. Πέραση τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. 20 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, μία αποχή. Merci beaucoup pour vos votes et toutes mes félicitations. ευχαριστούμε πολύ για την ψήφο σα και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια την κυρία Κατρίν Γκρέζ. Nous allons maintenant passer να περάσουμε τώρα στο σημείο 11 της ημερικής διάταξης. Il pas lui Σημείο 11 της ημερικής διάταξης αφορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Αλίας στην περιοχή του Ειρηνικού. Ο κύριος Πόγκα είναι ο εισηγητής. Μήπως ε, κάποιος τον ε, αντικαθιστά, η κυρία Στρίφλερ. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να σας ε, ζητήσω να κάνετε ησυχία σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Πόγκα μου ανέθεσε να παρουσιάσω το έργο του γιατί δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα το πρωί. Έτσι λοιπόν αντικαθιστώ τον κύριο Πόγκα ο οποίος ε, σας λέει το εξής. Θα σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που ε, εκπώνησα για τη ε, καθολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ελίας, στην περιοχή του Ειρηνικού. Καθώς είναι μεγάλο το θέμα και καθώς είμαστε περιορισμένοι στους 1500 χαρακτήρες, επικεντρώθηκα στις νήσους του Νότιου Ειρηνικού που συμμετέχουν στη Συμφωνία Κοτανού. Στην περιοχή του Ειρηνικού έχουμε 15 κράτη και που έχουν ε, ειδικέ σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου ο τομέα της Αλία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επιστηστική ασφάλεια και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Εγώ ήθελα να υπογραμμίσω πέντε στοιχεία. Καταρχήν, ότι είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε την απέτηση για τη συνοχή των πολιτικών της Ένωσης με τους ε, στόχους ε, της ανάπτυξης Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δράσεις της Ελίας στον ελληνικό εξασφαλίζουν αηφόρο βιώσιμη εκμετάλλευση των λευτικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή και να μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια περιφερειακή ε, στρατηγική. Είναι σημαντικό να προωθηθεί η θέσπιση ενό γενικού πλαισίου για την καλή διακυβέρνηση τη Ελία σε περιφερειακό επίπεδο στον ειρηνικό. Τρίτον, θέλω να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα να συντονιστούν οι διάφορες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή και κυρίως ε, την υποστήριξη στον τομέα της Ελίας ε, μέσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, του Μέσου και Συνεργασίας και του Πανδιατικού Μέσου για τον Ειρηνικό και των κονδύλιων προβλέπεται για το στήριξη στις χώρες ΑΚΕ. Επίσης, την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και αναρχισαλίας ε, και θα πρέπει να προσεγγιστεί και αυτό το θέμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει ρόλο στο θέμα αυτό. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι είναι αναγκαιότητα να ενημερώνεται η κοινωνία των πολιτών και οι επαγγελματικέ οργανώσεις όταν λαμβάνονται αποφάσεις για τον τομέα της αλίας. Είμαι στη διάθεσή σας και είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις σας για τη βελτίωση του κειμένου. Πρόσδεσμη μια κατάθεση τροπολογιών 12 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. 12 το μεσημέρι. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι που θα ήθελα να κάνουν σχόλια επί του θέματος αυτού. Διαφορετικά, να δώσω το λόγο στον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κύριε έρχεται το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομο θα είμαι. Τα βασικά σημεία τα ανέφερε η συνάδελφο Τρίφλερ. Υπενθυμίζουμε το θέμα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης που θεωρούμε προϋπόθεση για να μπορέσουμε να έχουμε συνοχή στις ε, συμφωνίες μας. Η παράνομη αλληλεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στο επίκεντρο ιδίω για αυτές τις περιοχές του ειρηνικού και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη για να τονίσουμε την υποστήριξή μας και για την κοινωνία των πολιτών. Είναι καλή έκθεση και θα ψηφίσουμε υπέρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέσπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την παρέμβαση των συναδέλφων. Νομίζω ότι όλοι θα υποστηρίξουμε την έκθεση. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις αλληλευτικές αυτές περιοχές και να μην τις αφήσουμε να θίγονται από την υπερεκμετάλλευση. Ε, είναι πολλοί στόλοι από Ασία, Αμερική ε, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους αλληλευτικούς πόρους και ιδίως ε, τον τόνο και πιστεύω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε εμείς τους πόρους, να τους εξασφαλίσουμε και για το μέλλον στο πλαίσιο της βιώσιμης πολιτικής. πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες μακροπρόθεσμα, όπως και σε άλλες αφρικανικές χώρες, να επιτραπεί η μακροπρόθεσμα βιώσιμη αλία και να μην υπάρχουν μεγάλα βιομηχανικά αλλιευτικά σκάφη. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και τα αποτελέσματα συνέργειας και να προστατεύσουμε και τις τοπικές περιοχές και τους ελευθερικούς πόρους ε, γενικότερα. Ως εταίρος ε, στο πλαίσιο ε, οικονομικών και ελευτικών συμφωνιών η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει αυτές τις περιοχές και να έχουμε τις καλύτερες δυνατές περιφερειακές ελευτικές συμφωνίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση και θα την υποστηρίξω. Ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βερόνικα Βάις ε, και ε, στην κυρία Ντεσούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ο κύριος Πόγκα στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, θέτει πολύ σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλία στο Ειρηνικό η Κομισιόν ε, μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τα περισσότερα από τα σημεία που υπάρχουν στο σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, Επίση, συμφωνούμε ότι η δατοκαλλιέργεια και η αελία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επιστημική ασφαλεία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των σχετικών κρατών ε, ε, και κυρίως των μικρών ισιωτικών ε, κρατών ε, στον ειρηνικό. Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην μακροπρόθεσμη αηφόρο ανάπτυξη και εκμετάλλευση των λευτικών πόρων στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να ωφεληθούν και μελλοντικέ γενιές. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει κοινή ευθύνη, υπάρχουν, υπάρχει ευθύνη και από τα παράκτια κράτη και από τα μικρά νησιωτικά κράτη να έρθουν σε συνεννόηση με τα άλλα μέρη που έχουν συμφέροντα στην περιοχή και αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ένα μικρό κομμάτι του στόλου της εκεί στον ειρηνικό και φυσικά εισάγει μεγάλες ποσότητες θαλασσινών στην Ευρωπαϊκή ε, αγορά. Επίσης, θα θέλω να σας αναφέρω ότι ε, οι αρμόδιες οργανώσεις, περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλίας ε, έχουν ε, συσταθεί δυνάμει του διεθνούς δικαίου και επίσης μαζί τους συνεργαζόμαστε για να καθολεμήσουμε την παράνομη δηλώτη ανεξέλεκτη αλία σε αυτές τις περιοχές. Έχω και μία ομάδα στη Μανίλα στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης της ε, των οργανώσεων διαχείρισης αλίας ε, το ειρηνικού που προσπαθούμε να προωθήσουμε μέτρα διατήρησης για τον τροπικό τόνο και για να καταπολεμήσουμε την παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία. Και να πω και δύο λόγια για την καλύτερη, οργάνωση, τον καλύτερο συντονισμό βρίσκεται στο κέντρο της ανακοίνωσης ε, της Κομισιόν για την ε, εξωτερική διάσταση της ελληνικής πολιτικής. Έχουμε δηλώσει την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε με άλλα τμήματα, κυρίως με το περιβάλλον, το εμπόριο, την έρευνα και την ανάπτυξη για να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση σε όλες τις δράσεις μας που στοχεύουν στον ειρηνικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 12 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 22 Ιανουαρίου του 2013. Τώρα, να περάσουμε στο σημείο 12 της ημερησίας διάταξης και στο σημείο 13. Θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο έκθεσης που αφορά την πρόθεση της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου. Η συγητής είναι ο κύριος Σβένσον. Και καθώς ο κύριος ε, Σβένσον πρέπει να παρουσιάσει και την γνωμοδότηση εμπόρου και ανάπτυξης βασισμένης επενδύσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και βασίζεται αυτή η γνωμοδότηση στο ίδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε προτείνω, αν συμφωνείτε κυρία Σβένσον, να δούμε αυτά τα δύο σημεία από κοινού. Για αυτή τη διπλή παρουσίαση θα υποδεχτούμε στο ιστορικό της Επιτροπής μας ε, τον κύριο Δενί Μπαρές από τη ΓΑΜΑ Δελτεμπορίου, τον κύριο Τζορζο Κόκκι ε, από τη ΓΑΜΑ Δελτα Ντεύκο και τον κύριο Μάρκ Μέσα, ο οποίος εκπροσωπεί την Κονκόρτ η εισηγήτρια για την έκθεση ΙΝΤΑ, η κυρία Σέφη, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση αυτή, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να περιβρεθεί. Χωρίς χρονοτριβή, να δώσω το λόγο στον κύριο Σβένσον για να μας ε, παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όπως ε, γνωρίζουν οι συνάδελφοι, έχουμε δύο παράλληλες εκθέσεις για το ίδιο ζήτημα εδώ. Η μία είναι έκθεση στην Επιτροπή ΔΕΒΕ και η άλλη είναι μια γνωμοδότηση για την ε, έκθεση ΣΑΙΦΗ για την ε, ΙΝΤΑ. Όπως ξέρετε και τα δύο αυτά εγγραφά θα είναι αλληλοσυμπληρωματικά. Εγώ ελπίζω ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικές ε, προοπτικές πάνω στο ίδιο θέμα και θα υπάρχει άλλο συμπλήρωμα των δύο επιτροπών. Η έκθεσή μου συζητήθηκε για πρώτη φορά στην ε, δική μας επιτροπή πριν ένα μήνα και προσπάθησα να τονίσω το ρόλο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην ε, πρόθεση της ανάπτυξης στις φτωχές χώρες αν ε, δηλαδή ε, υλοποιηθούν αυτά με υπεύθυνο τρόπο. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι το εμπόριο είναι μία από τις πιο σχετικές πολιτικές, ένα από τους πιο σχετικούς τομείς πολιτικής ε, για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ε, παγκοσμία ανάπτυξη. Αν η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής χρησιμοποιηθεί καλά, τα εργαλεία του εμπορίου μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στι φτωχέ χώρε από πολλέ αναπτυξιακέ πολιτικέ. Το σημαντικό είναι οι εμπορικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια των αναπτυσσόμενων χωρών να έχουν ω κύριο στόχο να εξυπηρετούν και να ενισχύουν τα αποτελέσματα των πολιτικών βοήθειας. Ε, αυτή είναι η κύρια προσέγγιση μου στις εκθέσεις μου. Εγώ σε μία παράγραφο αναφέρομαι στις πρωτοβουλίες βοήθειας που έχουν ως στόχο να αυξήσουν την ικανότητα του εμπορίου στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό αποκαλείται Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο. Ίσως ε, να επαναλαμβάνω κάποια θέματα, αλλά είναι σημαντικό εμείς να βάλουμε τα δυνατά μας για να αυξήσουμε την ικανότητα των ε, φτωχών χωρών να μπορούν να διαχειρίζονται το διεθνές εμπόριο και να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο σύστημα και να κερδίζουν χρήματα από αυτό. Αυτό χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες, αν να ε, αποτελέσουν ε, ε, επιτυχές τμήμα της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει οι φτωχές χώρες να ενταχθούν και να αποτελέσουν τμήμα του διεθνούς εμπορίου και όχι να παγιδευτούν στο ρόλο των παραγωγών πρώτων υλών και μόνο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα κύρια στοιχεία για να μειώσουν την εξάρτησή του από τη βοήθεια και να μειωθεί η ανέχεια. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εμπορικές συμφωνίες, είναι απολύτως θεμελιώδες για τις αναπτυσσόμενες χώρες να μπουν σε αυτές τις συμφωνίες, να συνάψουν τέτοιες συμφωνίες. Νομίζω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τι αναπτυσσόμενες χώρε να μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιε τι είναι σωστό για αυτέ και ποιε συμφωνίε θέλουν να προσυπογράψουν ή ποιε συμφωνίε δεν θέλουν να συνάψουν. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζουμε. Βασιζόμαστε στο ότι όλοι έχουν ε, ίση αξία. Έτσι λοιπόν, ε, με τον ίδιο σεβασμό θα πρέπει να συναντήσουμε στις διαπραγματεύσεις και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες θυσίες στις διαπραγματεύσεις μας. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης πρέπει να ενθαρρύνουμε τους συνομιλητές μας να λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον όλου του πληθυσμού και ολόκληρη τη χώρα όταν διαπραγματεύονται. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά όσοι εκπροσωπούν μια χώρα και έχουν την εντολή τη διαπραγματευτική εκ μέρου τη χώρα αυτή, πολύ συχνά σκέφτονται μόνο τα συμφέροντα μια κάποια ελίτ. Φυσικά τελικά η ίδια η χώρα είναι αυτή που θα πρέπει να τα ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα. Όμω νομίζω εμεί ότι από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνουμε κάτι, να ερθαρρύνουμε τι χώρε να έχουν ε, μια πιο ε, ολοκληρωμένη διαδικασία ω προ τι διαπραγματεύσει. Τώρα, για να μιλήσουμε για το εμπόριο. Ε, όσοι ζούμε σε αναπτυγμένες χώρες έχουμε την ευθύνη να είμαστε σίγουροι ότι δεν ε, συνεισφέρουμε ε, σε χώρες όπου υπάρχει πείνα να χρησιμοποιείται η οικονομική γη για κάτι άλλο πέρα από τις καλλιέργειες ε, για να τραφεί ο τοπικός πληθυσμός. Εγώ καταδικάζω ότι η γη πολλές φορές χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αν θέλουμε να επιτύχουν οι χώρες αυτές στο διεθνές εμπόριο, εμείς ε, μαζί με τις προσπάθειες που θα καταβαλούμε για να ενταχθούν καλύτερα οι φτωχές χώρες στο διεθνές εμπόριο πρέπει να προωθήσουμε πέραν αυτού την ανάπτυξη και την επασχόληση στους τομείς όπου είναι ενεργοί οι πιο φτωχοί. Όπως ε, γνωρίζετε, οι βουλευτές μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις. Εγώ δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω στην έκθεση όλα όσα ήθελα και θα καταθέσω μια σειρά τροπολογιών στην έκθεσή μου και εγώ ίδιος. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος πολλά περισσότερα σε σχέση με τις ευκαιρίες και τα προβλήματα που ε, μπορεί να παρουσιάσει η απελευθέρωση του εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια, ο στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας ε, και ε, βελτίωση του επίπεδου ζωή στι χώρε αυτέ. Όμω πρέπει να καταπολεμηθούν και αρνητικέ συνέπειε, όπω παραδείγματο χάρη η απώλεια φορολογικών και τελωνιακών εσόδων. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα έχει να κάνει με τις ευκαιρίες να βελτιώσουμε ε, το πώς ε, λειτουργεί, ποιες είναι οι συνθήκες στις εξωτερικές βιομηχανίες. Χαίρομαι που έχουμε εδώ και πρόσωπο από την Concord. Ε, σίγουρα και εσείς έχετε πάρα πολύ ωραίες ιδέες να μας αναφέρετε εδώ και ανυπομονώ να ακούσω και τις ε, απόψεις των εκπροσώπων της Κομισιόν και από την Concord αλλά και των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σβένσον και δίνω τώρα το λόγο στην Επιτροπή που εκπροσωπείται τον κύριο Ντενί Μπαχέσου και μετά θα δώσω το λόγο και στους υπολείπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. είμαι Μπερές, δουλεύω για την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και έχω ασχοληθεί με την προετοιμασία αυτή τη έκθεση μαζί με τον φίλο Τζόρτζιο από την ΑΔΕΦΚΟ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Σπένσον, για την έκθεσή του. Χαιρετίζουμε τη σύγκληση των απόψεων σε πολλά σημαντικά θέματα, όπως τη σημασία ε, του εμπορίου, τη σημασία της λειτουργίας των εσωτερικών και περιφερειακών αγορών, καθώς ε, και πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η διακυβέρνηση και το θέμα της οικειοποίησης αυτών ε, των στόχων από τους ίδιους τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς αυτό. Θέλω να κάνω και κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχήν να πω ότι από τη δική μας οπτική γωνία θεωρούμε ότι αυτή η νέα ανακοίνωση δημιουργεί ένα όραμα για το μέλλον και δίνει σαφείς ε, κατευθύνσεις για την ε, ε, εμπορική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξη. Ξεκινώ με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τα έχουμε στην παράγραφο Β. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου ήδη διεξάγεται στο πλαίσιο των ε, στόχων ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και αυτό διασφαλίζει και τα, ε, την προσοχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και αυτό ισχύει για το σύνολο της εμπορικής πολιτικής που περιλαμβάνει και το εμπόριο και την ανάπτυξη βέβαια. Άκουσα τον εισηγητή και βλέπω και την παράγραφο σίγμα Και υπενθυμίζω ότι υπάρχει τώρα ένα αντίστοιχο σύστημα. Θα συνεχίσει η Επιτροπή να είναι πολύ ευέλικτη σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι δεν υπάρχει ε, αμφιβολία ότι τους εταίρους μας τους μεταχειριζόμεθα ως απόλυτα ισότιμους εταίρους δεν πιέζουμε κανένα να κάνει οτιδήποτε. Και τελικά πιστεύω ότι για να φτάσουν σε τελική φάση αυτές οι διαπραγματεύσεις χρειάζεται η πολιτική απόφαση για να καταλήξουν κάπου αυτές τις συμφωνίες. Ίσως αυτό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τις σχετικές παραγράφους GI και πρέπει να πούμε ότι ε, το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα ανοίξει νέες ε, εξαγωγικές ε, προοπτικές. οι προτιμήσει απευθύνονται στι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και γι' αυτό πιστεύω ότι θα προκύψουν ευκαιρίε υπό δύο μορφές. Θα υπάρχει λιγότερο ανταγωνισμό σε τομεί όπου οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες είναι ήδη παραγωγή και δεύτερον οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες έχουν τώρα την ευκαιρία της διαφοροποίησης ώστε να επωφεληθούν από την μείωση των δασμών σε τομείς όπου βρίσκονταν υπό την ανταγωνιστική πίεση των πλούσιων αναπτυγμένων χωρών. Έχει γίνει λεπτομερής ε, εκτίμηση επιπτώσεων ε, στο πλαίσιο της ε, μεταρρύθμισης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και όλα αυτά τα θέματα έχουν καταγραφεί. Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τους πόρους, και την κατάρα των πόρων όπως ε, ονομάζεται ιδίως για την υποσαχάριο Αφρική ε, εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αυτό εποφελούνται οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από την ευρωπαϊκή αγορά για όλα τα προϊόντα τους εκτός από τα όπλα και τους, εξοπλισμούς βέβαια δεν δίδεται πλεονέκτημα στις πρώτες χείλε έναντι των μεταποιημένων προϊόντων, αλλά δεν δημιουργείται εδώ ε, κανένα μειονέκτημα και δεν υπάρχει και περιορισμός στις εισαγωγές. Τηρούμε βέβαια τις συμφωνίες οτιδήποτε εκτός από όπλα ε, και όλους τους κανόνες που έχουν σχέση με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Πάντως οι κανόνες είναι απλοί για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να υποφεληθούν από αυτά τα συστήματα με τρόπο ώστε να προωθηθεί το εμπόριό τους. Ένα σημαντικό θέμα είναι στην παράγραφο ΙΓ που αφορά την αρπαγή γης. Εδώ η Επιτροπή πιστεύει ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα και να δημιουργηθούν ευκαιρίε απασχόληση και να μειωθεί η φτώχεια. Παρ' όλα αυτά, θέλω να διευκρινίσω ότι θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό τέτοιου είδου επενδύσει να γίνονται με τρόπο υπεύθυνο και μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Γι' αυτό και υποστηρίζουμε εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες για τον προσδιορισμό των αρχών και κώδικα δικαιολογίας για τις επενδύσεις σε γεωργική γη. Υπάρχει και το θέμα των στόχων στην παράγραφο 10. Εδώ διαφωνούμε με αυτή την έννοια των αναπτυξιακών στόχων μέσα σε μια συμφωνία για την ανάπτυξη του εμπορίου. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα βοηθήσουμε ε, στην παρακολούθηση και στην αναθεώρηση και θα γίνει αναθεώρηση των συμφωνιών μαζί με τους εταίρους μας, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Θα χρειαστεί ορισμός δικτών από όλους τους εταίρους από κοινού, όπου αυτό είναι απαραίτητο, αλλά πιστεύω ότι δεν πρέπει μέσα στη συμφωνία να ορίζονται δείκτες γιατί ίσως να χρειάζεται μια προσαρμογή τους με το πέρασμα του χρόνου για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον, παραδείγματο χάρη, και παρότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται στις ε, αλλαγές ε, των ε, ε, στόχων δεν πρέπει να είναι αυτόματες αυτές οι προσαρμογές γιατί αν γίνονται αυτόματες προσαρμογές αυτό θα είναι κατά του αρχικού στόχου που έχουμε του να προωθήσουμε βιώσιμες αλλαγές. Τώρα όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη παραγράφους 15 και 16 συμφωνούμε απολύτως με τις γενικές αρχές της εταιρική ευθύνη και ο εθελοντικός χαρακτήρας είναι πάρα πολύ σημαντικός για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση απόδοση. Παράγραφος 19 για τη διαδικασία Kimberley. Ε, όπως γνωρίζετε διαφωνούμε. Εδώ έχουμε μια αρνητική αξιολόγηση για τη διαδικασία Kimberley. Τα διαμάντια από περιοχές σύγκρουσης αποτελούν 1% του διεθνούς εμπορίου σε διαμάντια Αντίθετα, τη δεκαετία του 90 ε, είχαμε αντίστοιχε εκτιμήσεις ε, του επίπεδου 15%. Η συμφωνία λοιπόν Κίμπερλι βοήθησε να σταθεροποιηθούν χώρες. Έχουμε μια πολύ πιο θετική αντιμετώπιση λοιπόν της διαδικασίας Κίμπερλι εμείς σε σχέση με τις ελλείψεις που επισημαίνονται εδώ. Στις παραγράφους 21 και 22 για την ασφάλεια των τροφίμων Έχουμε λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Στις 17 Οκτωβρίου υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο μία πρόταση για την μείωση της ε, συνολικής παγκόσμιας επιφάνειας για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και για τα εισαγόμενα βιοκαύσιμα. Και σύμφωνα με την πρόταση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ένα περιορισμό στο 5% που ε, αντιστοιχεί στην τωρινή κατανάλωση τηρώντας ε, το στόχο του 5% για ανανεώσιμη ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα θα πρέπει να έρθουν από βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Ο στόχος της πρότασης είναι να υποκινήσουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων δεύτερης γενιάς που δεν θα είναι από ε, επισητιστικά προϊόντα, θα μπορούσαν να είναι από άχυρο ή από απόβλητα. Τώρα, ο Τζόρτζιον πώς θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο για να συμπληρώσω την παρουσίαση του συναδέλφου. Θέλω και εγώ να μιλήσω για ορισμένα σημεία στα οποία πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Στο σημείο 5 για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη σε πολλούς τομείς μπορεί να βελτιώσει ε, τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της φτώχειας, εφόσον τα ωφέλη από την ανάπτυξη κατανέμονται αποτελεσματικά. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεση του εισηγητού, αλλά εδώ το κείμενο δίνει την εντύπωση ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη, ιδιαίτερα στους τομείς ε, όπου δραστηριοποιούνται οι άποροι άνθρωποι. Εγώ δεν θα το εξέφραζα έτσι, γιατί υπάρχουν τομείς όπως η ανάπτυξη της υπαίθρου, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση απόρων, ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες, και θα μπορούσε να είναι αποδοτικέ οι επενδύσει, ε, Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου η ανάπτυξη θα μπορούσε να βοηθήσει την μείωση της φτώχειας. Εγώ λοιπόν δεν θα το εξέφραζα τόσο κατηγορηματικά. Αυτή είναι η πρότασή μου για την παράγραφο 5. Στην παράγραφο 13 που αφορά τα μέσα που έχουμε για τη βοήθεια για το εμπόριο, συμφωνούμε απολύτως με το περιεχόμενο της παραγράφου, Πιστεύουμε επίσης ότι σήμερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους δωρητές, η κατάσταση είναι τέτοια που δεν περιορίζουμε τη βοήθεια για το εμπόριο. Πρέπει να πούμε εξάλλου ότι η βοήθεια για το εμπόριο που χορηγούμε εμείς είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίω. Και δεν περιορίζουμε αυτή τη βοήθεια στην υποστήριξη του εμπορίου μεταξύ αναπτυγμένων χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά πρόγραμμα. Την περασμένη εβδομάδα καταμετρήσαμε πάνω από 100 προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρο τον κόσμο στο πλαίσιο της βοήθειας για το εμπόριο. Δηλαδή δεν διαφοροποιούμε τις περιπτώσεις που έχουμε εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυσσομένων χωρών ή εμπόριο νότου-νότου ή μεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Και στην επόμενη παράγραφο, στην παράγραφο 14, Συμφωνούμε με τους στόχους της παραγράφου σε γενικές γραμμές, αλλά η διαφοροποίηση πρέπει να πούμε ότι απαιτεί επενδύσεις που εξαρτάται κατά πολύ από το επιχειρηματικό περιβάλλον και την οικονομική διακυβέρνηση. Υπάρχει δηλαδή κάποιο όριο στο τι μπορούν να κάνουν οι εξωτερικοί δωρητές. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή και πάλι ότι φέρουν ευθύνη και οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες που πρέπει να αναλάβουν τη δική τους αναπτυξιακή πολιτική. Εμείς ήδη βοηθούμε αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά δεν υποκαθιστούμε την πολιτική βούληση στις ίδιες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μετά, στην παράγραφο 17, σε σχέση με τους φορολογικούς παραδείσους, η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι ένας εύκολος τομέας, στον οποίο θα μπορέσουμε εύκολα να έχουμε αυτά αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε ε, να εκτιμούμε ιδιαίτερα την βοήθεια που παρέχει το Κοινοβούλιο στο διάλογο με τα κράτη-μέλη, διότι γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών. Ήθελα όμως να καταγραφεί η δράση η οποία ήδη διεξάγεται σε αυτό τον τομέα. Για τη διαδικασία Κίμπερλι ήδη είπε ο συνάδελφος ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Για την παράγραφο 21 και την παράγραφο 22 για την ασφάλεια των τροφίμων θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Ίσως θα ήταν καλύτερα κάπως να διευκρινίσουμε το μήνυμα που θέλουμε να βγει προς τα έξω ίσως υπάρξει παρανόηση ότι η ασφάλεια των τροφίμων εξαρτάται πάντοτε από την κατατόπους παραγωγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένα χρονικά σημεία και ορισμένες περιφέρειες μπορεί αυτό να ισχύει. Αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές που γνωρίζουν οι οικονομολόγοι, δηλαδή ότι η ασφάλεια των τροφίμων εξαρτάται και από τη δυνατότητα αγοράς τροφίμων στην αγορά. Δηλαδή όχι μόνο από την τοπική παραγωγή, από την εθνική παραγωγή, αλλά και από την ικανότητα αγοράς τροφίμων τα οποία βρίσκονται διαθέσιμα κάπου αλλού. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να επαναλάβω ότι γενικά συμφωνούμε με τις βασικές γραμμές του κειμένου. Ευχαριστώ. Κονκόρντα. Ο κ. Μαρκ Μέσεκ προσωπεί την Κονκόρντα. Thank uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που επιτρέπετε στην Concord να λάβει το λόγο εδώ. Όπως ξέρετε η Concord ε, είναι η λογική φορέας ε, ομπρέλες ε, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Ευρώπη και εγώ εργάζομαι ως σύμβουλο στη Βελγική Πλατφόρμα Θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ πλούσια η έκθεση με πολλές νέε απαντήσεις και αναφέρονται πάρα πολλά πράγματα που εμεί θεωρούμε σημαντικά, όπως παραδείγματο το ότι επιμένεται στην ισότητα των δύο φίλων στην καλή διακυβέρνηση, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική συμμετοχή κτλ. Υπάρχουν ε, δύο στοιχεία νομίζω που λείπουν και βεβαίως ε, θα μπορούσα να συζητήσω και με την Επιτροπή για τα θέματα που ακούστηκαν, όμως ε, σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις της Κομισιόν, δεν ε, είναι κακό να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα ακόμη και αν εφαρμόζονται ήδη από την Κομισιόν. Είναι σημαντικό επίση λοιπόν να τονίζουμε και συμφωνεί το Κοινοβούλιο ότι κάποια πράγματα πρέπει να πηγαίνουν προ συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά μα λείπουν τα δύο εξή. Καταρχήν, είναι αλήθεια ότι η ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής, μίσου της στόχια, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Αλλά αν δείτε την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και αν δείτε συγκεκριμένα το άλλο έγγραφο για την ανάπτυξη του εμπορίου και τις παγκόσμιες υποθέσεις, αυτό το έγγραφο καθορίζει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Εμπόριο, όχι το έγγραφο που συζητείτε εδώ. Αν δείτε λοιπόν εκείνο το έγγραφο, θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική καταρχήν ε, έχει ως στόχο να πετύχει επιθετικά και αμυντικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αμυντική και εμπορική πολιτική που προσπαθεί να πετύχει πρόσβαση στην αγορά, όσο δυνατόν περισσότερο παγκοσμίω και να διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκά προϊόντα και επενδυτέ να μπορούν να μπουν σε αγορέ, ότι οι ευρωπαίοι επενδυτέ θα μπορούν να είναι παρόντε σε αγορέ και θα υποφελούνται από ιδιαίτερη εθνική μεταχείριση. Δηλαδή, ουσιαστικά να λάβουν ε, ένα ικανό μερίδιο της ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Πρόκειται λοιπόν για μια επιθετική πολιτική και αυτό που τονίζουμε εμείς και υπάρχει και στην έκδοση είναι ότι ε, και η οικειοποίηση είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει και οι αναπτυσσόμενες χώρες να καταρτήσουν τα δικά τους αναπτυξιακά σχέδια και να εντάξουν το εμπόριο στα σχέδια αυτά και να εργαστούν για αυτό το στόχο. Και αυτό που βλέπουμε στην εμπορική πολιτική είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει φυσικά στην επίτευξη των δικών της συμφερόντων που δεν ταιριάζουν απαραίτητα με τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών. Ως αποτέλεσμα, πολύ συχνά στις εμπορικές διαπραγματεύσεις βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση ζητά απελευθέρωση εκεί όπου ε, δεν σκόπευαν να πάνε οι αναπτυσσόμενε χώρε και για ταχύτητα που δεν σκόπευαν να έχουν οι αναπτυσσόμενε χώρε. Έτσι λοιπόν υπάρχουν συνεχεί αναντιστοιχίε και γι' αυτά πολλά από τα μέλη τη Concord εργάζονται επί εξτρατιών για να διασφαλίσουν ότι τα επιθετικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάπω υποβαθμίζονται, αποδυναμώνονται. Αναφέρθηκε η ανάγκη να γίνουν θυσίε από την Ευρώπη, να ανοιχτεί λίγο περισσότερο νομίζω νομίζω ότι το πιο προβληματικό θέμα με την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι ότι είναι επιθετική και αν ε, πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μειώσει τις φιλοδοξίες της προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεύτερον, και σχετίζεται με το πρώτο, αν δείτε τη βοήθεια για το εμπόριο, Ξέρετε ότι από το 2005 στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε σημαντικά και είναι στην πρώτη θέση η Ευρώπη στον τομέα αυτό. Οι περισσότερε αξιολογήσει ε, που είδαμε για τη βοήθεια για το εμπόριο και πρόσφατα λάβε χώρα και μια συνδιάσκεψη στη Γενέβη. Οι ε, περισσότερε λοιπόν από τι αξιολογήσει επαναλαμβάνουν ότι συχνά υπάρχει ένα αντιστοιχεία μεταξύ τη αξιολόγηση των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από του δωρητέ. Και πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι δεσμεύσει από του δωρητέ ε, πηγαίνουν σε κλάδου που ενδιαφέρουν του δωρητέ. Παραδείγματο χάρη ένα καλό παράδειγμα είναι το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το PAPET, που θέλει η Δυτική Αφρική να ε, το συνδέσει με τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Εκεί ε, βλέπετε τι ανάγκες έχει κάθε χώρα σε κάθε τομέα και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε από την άλλη πλευρά τι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, ε, κάποιες χώρες ε, που τις ευνοούν δωρητές ε, και βρέπετε ότι σε πολλούς τομείς δεν υπάρχει πρόθεση αυτών των μέσων κάποιες χώρες. Στην... Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει αναντιστοιχεία και φυσικά αυτό έχει να κάνει με το ότι όταν χορηγείται η βοήθεια για το εμπόριο, οι διεθνείς δωρητές προσπαθούν επίσης να διευκολύνουν και την υλοποίηση των δικών τους στόχων. Στο παράδειγμα της Κίνας ε, υπάρχει παραδείγματος χάρη ε, μία παραχώρηση για ένα ορυχείο και τελικά φτιάχνουν ε, και έναν αυτοκινητόδρομο από το ρηχείο μέχρι τη θάλασσα. Αυτό τους διευκολύνει και για τα δικά τους σχέδια για να μεταφέρουν τις πρώτες ύλες. Επομένως, ε, λοιπόν, ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέτει ως προτεραιότητα σε πρώτη θέση τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Για να κλείσω. Αναφερθήκε και η Κομισιόν ε, σε δύο θέματα, τη συμφωνίες οικονομικές και εταιρικές σχέσεις ε, και στο ΕΣΠΗ. Να σας πω ότι η μεταρρύθμιση ε, του GSP δεν σημαίνει ότι θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Εμείς έχουμε κάποιες αντιρρήσεις, έχουμε υποβάλει πολλές συναλλακτικές προτάσεις και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν και εμεί πιστεύουμε ότι το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων όπω έχει αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο γενναιόδωρο από ό,τι πριν και αν δείτε τι συζητήσει που έλαβαν χώρα όταν προσαρμόστηκε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα δείτε ότι επίσης υπήρξαν εκεί και επιθετικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα υπήρξαν και προτάσεις να ε, ασκηθεί πίεση σε κάποιες χώρες αναπτυσσόμενες για να διαπραγματευτούν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Έτσι λοιπόν, το σχάρι, αν θέτουμε προθεσμίες, αυτό δημιουργεί πίεση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, να, προτιμούμε να, αποσύρουμε, προσπαθούμε να αποσύρουμε προτιμήσεις και αυτό ασκεί πιέσεις και οθούνται οι χώρες προς κάποιες κατευθύνσεις. Και τώρα για τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρική σχέσης. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι ευέλικτη η Κομισιόν, ε, είναι μάλιστα αυστηρή και γι' αυτό καθυστερούν τόσο πολύ αυτέ οι διαπραγματεύσει. Έτσι λοιπόν και πάλι παροτρύνουμε την Κομισιόν να είναι πιο ευέλικτη από όσο είναι σήμερα. Merci. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μίτσελ τώρα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή και για τις ε, προσπαθίες σας και το χρόνο σας. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για το είπε και τις απαντήσεις της Concord. Εγώ θα ήθελα να θέσω κάποια ζητήματα για την αναπτυξιακή πολιτική και το πώς ε, θα προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω του εμπορίου. Γιατί πολλοί εδώ και πολλά χρόνια, βλέπω και τον κύριο Ντεβέδο, έχουν ε, παρουσιάσει κάποια θέματα που αφορούν την αύξηση της ε, ικανότητας εμπορίου σε αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να μας πει η Κομισιόν τι έκανε, παραδείγματος χάρη, για να ενθαρρύνει την ε, ιδιοκτησία, αποκτήση ιδιοκτησίες. Παραδείγματος χάρη, Πώς μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους ε, την ικανότητα για το εμπόριο και να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν ε, το χάρη, τι γίνεται ακριβώ με την ε, ιδιοκτησία, δηλαδή πώ βοηθάει η Κομισιόν τους πολίτε να δημιουργήσουν εμπόριο. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα, να δούμε τη δική μου χώρα, η Ιρλανδία διαιρέθηκε δηλαδή γιατί κάποιοι, ε, σε κάποιους δόθηκαν μικρά αγροτεμάχια και μπορέσαμε κατόπιν να τα εκμεταλλευτούμε και να ε, δημιουργήσουμε βιομηχανία. Επίση επίσης, να σας πω ότι πριν ε, δύο εβδομάδες ε, στο Στρασβούργο συζητήσαμε το ότι παραδείγματος χάρη κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους για να αναπτύξουν το πεζικό σύστημα και όπου δεν υπάρχει. Και ξέρω ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όπως και στην Αφρική. Όταν επισκέφθηκα αυτές τις χώρες, ξέρω ότι οι περισσότερες ε, από τους νέους μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα το κινητό από μένα. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια ευκαιρία, χρησιμοποιούμε τέτοιε ευκαιρίε για να οικοδομήσουμε παραδείγματο χάρη, ένα τραπεζικό σύστημα εκεί όπου δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Και επίσης ε, το θέμα των ε, ε συστημάτων ε, διασφάλισης των σοδιών, παραδείγματο χάρη. Πώς μπορούμε να δώσουμε ε, στους πολίτες ε, ε, και την αίσθηση να προωθήσουμε κάποιο σύστημα στο οποίο θα λένε ότι δεν πρέπει να έχουμε 12-15 παιδιά επίσης για τους ανθρώπους με εμπειρίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο Αναφέρεται η έκθεση συγκεκριμένα και στο να προωθηθεί η ανάπτυξη μέσω του εμπορίου, επενδύοντας τις ευκαιρίες για τις γυναίκες, που γενικά έχουν υψηλές αποδόσεις σε ό,τι αφορά την οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη, σε ό,τι αφορά τώρα στην εμπορική μας πολιτική, για να δώσουμε την ικανότητα στους ανθρώπους να εμπορεύονται. Τι πιστεύει η Κομισιόν, ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων με και των γυναικών και μπορείτε να τους δώσετε την ευκαιρία και αυτοί να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε και να αναπτύξουμε αυτό το επιχειρηματικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ. Merci. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μένα θα προσφέρω το λόγο. Ευχαριστώ τον κύριο Σβέντσον για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Μιλήσατε για φορολογικούς παραδείσους ε, και αναφερθήκατε και στις πρώτες ύλε. αλλά και στο ότι οι εταιρείες ε, θα πρέπει να είναι υπεύθυνε. Εγώ νομίζω ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα πρέπει να είναι δεσμευτική. Δεν μπορεί να είναι προαιρετική και να εξαρτάται από την ίδια την εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, στην έκθεση αυτή υπάρχουν κάποια πράγματα που λείπουν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τα τέλη, τους δασμούς τελωνιακούς. Δεν μπορούμε αυτούς τους δασμούς τελωνιακούς να τους μειώσουμε χωρίς να υποστούμε ζημιά σε αυτή την αναπτυγμένη οικονομία αυτά, αυτοί οι δασμοί είναι ορισμένα μονάδες ε, στα έσοδα 5-10 και στο Αφγανιστάν είναι 40% του προπολογισμού. Στη Μαδαγασκάρη είναι 50% του προπολογισμού. Άρα λοιπόν το να αφαιρέσουμε αυτά τα εμπόδια σημαίνει ότι έτσι απότομα οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν δυσκολίες και το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Σημαντικότατο λοιπόν είναι για μας ε, οι χώρες αυτές να μπορέσουν να προσαρμοστούν ε, χωρίς τους τελωνιακούς δασμούς να τους αφαιρέσουν, να τους ε, καταργήσουν έτσι απότομα και γι' αυτό να υπάρχει μια κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης ε, υποχρεωτική δεσμευτική. Θέλουμε να αποφύγουμε αυτό που είδαμε πάνω στην Ιγυρία ότι το περιβάλλον καταστράφηκε από πολυεθνικές οι οποίες ε, χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται ε, στο, τις ε, παραγωγικές πηγές όπως και στο Νίγερα, την Αγέβα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνη η μητρική εταιρεία για όλες τις καταστροφές λόγω της εξόριξης πρώτων υλών και της εκμετάλλευσής τους. Αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις αυτές να συμμετάσχουν στην τοπική ανάπτυξη και όχι όπως το διαπιστώσαμε τα τελευταία 40 χρόνια που κουρσεύουν τους πόρους, δεν πληρώνουν τίποτα, ούτε φόρους ούτε τίποτα και μετά φεύγουν, εγκαταλείπουν τη χώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς τώρα έχει το λόγο. Ναι, και εγώ θα ήθελα ευχαριστήσω τον κ. Βάσεν ε, για την λεπτομερή πραγματικά έκθεσή του που επιμένει σε διάφορους τομείς που μας απασχολούν σίγουρα από όταν ξεκινήσαμε να ασχοληθούμε με παρόμοιες εμπορικές υποθέσεις. Ε, θέλω να δείξω το εξής εγώ να μην υποτιμάμε την δύναμη του εμπορίου και να μην υπερτιμούμε το πώς μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση για τα φτωχά στρώματα του Εδώ ε, όλα αυτά που είπαμε πριν ε, δεν ε, λύνουν το πρόβλημα, αλλά είναι συνοδευτικά μέτρα και για να μπορέσουν όσο γίνεται να ωφεληθούν οι πληθυσμοί από τα θετικά αυτά σημεία. Τι θέλω λοιπόν να πω αποσιωπούμε ιδιαίτερα την άτυπη οικονομία, στην πούμε έτσι, ε, αφρικανικές χώρες. Ε, είναι το προκαταρτικό στάδιο. Πρόκειται για μια εισαγωγή πριν ε, την επίσημη οικονομία αυτή, η άτυπη οικονομία είναι αυτή που ξεκινάνε από το μηδέν να περάσουν από ένα διάμεσο στέδιο, να μάθουν, να διδαχτούν, να εξοικονομήσουν κάτι και να μπορέσουν ε, να δημιουργήσουν κάτι που να επαρκέσει για τις ανάγκες τους. Και αυτή η άτυπη οικονομία απειλείται όμως από το εμπόριο και από το διεθνές εμπόριο. Σημαίνει ότι διάφορα προϊόντα έχουν πολύ χαμηλές τιμές ε, που πουλούνται εκεί σε αυτή την άτυπη οικονομία, στα πλαίσια της, ε, από χώρες ε, ιδιαίτερα παρούσες ε, στην Αφρική όπως την Κίνα και την Ινδία και όσοι πήγατε σε αφρικανικές χώρες ε, βλέπετε στους δρόμους χιλιόμετρα ολόκληρα με προϊόντα που πουλούν μέσω της, αυτού του εμπορίου τους περαστικούς τα πολλούν αυτά τα προϊόντα και αυτά τα προϊόντα είναι προέλευσης όχι αφρικανικής. Και αυτά δεν έχουν να κάνουν με το dumping το κοινωνικό, αλλά το νομισματικό dumping. Και εδώ δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανένα στο δικαστήριο, ε, στη Γενέβη, αλλά έχει τα ίδια αποτελέσματα γιατί ε, δεν αφήνει για πολλά χρόνια να επιτευχθεί μια ανάπτυξη. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Είχαμε και μια διάσκεψη ανάμεσα στην Κίνα και στις ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ τρία λεπτά όλα και όλα εξήγησαν το πρόβλημα οι Ευρωπαίοι και μια βία, ας την πούμε έτσι απάντηση από την άλλη μεριά γι' αυτό δεν συνεχίστηκε η συζήτηση δεν είναι με τη σιωπή που θα μπορούσε κανείς να λύσει παρόμοια θέματα. Έτσι χρειάζεται να τα δούμε, να τα σκεφτούμε και να λύσουμε για καλύτερες μορφές προστασίας των αφρικανικών χωρών. Το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Θα πρέπει μια στρατηγική να αναπτύξουμε για να το πετύχουμε, έτσι. Και καθόλου μα καθόλου εύκολο δεν θα είναι. Η πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική σε αυτήν την περίπτωση. Ένα ακόμα στοιχείο δε Υπάρχουν συνέπειες ε, αρκετά σημαντικές στην Αφρική. Μέση ανάπτυξη της τάξης του 5% πάνω από το ποστό Πραγματική ανάπτυξη. Μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι στο σύνολό της η Αφρική μακροοικονομικά μιλάω, έτσι. Αντιστάθηκε περισσότερο στην κρίση από οποιονδήποτε άλλον. Δεν ξέρω. Σωστά ή όχι σωστά αλλά έχει παρακάμψει την κρίση του χρέους. Υπάρχουν δυνατότητες και το αφρικανικό χρέος ε, είναι εσωτερικής φύσεως. Ε, υπάρχουν εξελίξεις ιδιαίτερα θετικές που θα πρέπει να ενθαρρύνουμε. Επίσης θα πρέπει να ρωτηθούμε το εξής. Το εμπόριο της Αφρικής ε, πώς συμμετέχει στον υπόλοιπο κόσμο καθόλου σχεδόν, ενώ η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ισχυρότερο ρυθμό. Και νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερε δυνατότητε. Αρχίζει κανεί να την εκμεταλλεύεται. Είναι το ενδοαφρικανικό εμπόριο ανάμεσα σε διάφορε περιοχέ τη Αφρική. Λυπάμαι πραγματικά γιατί με την εταιρική αυτή σχέση με τι συμφωνίε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όσο γρήγορα επιθυμούμε. Και αυτό οφείλεται σε ένα πρόβλημα όλου μηχανισμού, στο μηχανισμό που ίσχυσε εδώ και μερικά χρόνια και τα βάλαμε όλα στους ώμους του αρμόδιου επιτρόπου για το εμπόριο και αφήσαμε στην άκρη τον επίτροπο για την ανάπτυξη ενώ συμφωνούν όλοι ότι οι σχετικές συμφωνίες θα πρέπει να αφορούν όλες τις διαστάσεις του προβλήματος, διαφορετικά θα τα πετύχουμε. Όλα λοιπόν με την προστασία της εβέστη ακόμα ευαίσθητης ευάλωτης αγοράς και το συμφέρον μας είναι να, ε, να εμπνευστούμε από το μια κούλπα του Κλίντον στη Γερουσία την Αμερικανική που είπε για την ε, υποχώρηση της αγροτικής οικονομίας της ΑΕΤΙΣ και είπε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη του. Ποια ήταν αυτή η ευθύνη ότι εκείνος ε, θανάτωσε την γεωργία της ΑΕΤΙΣ ε, γιατί δεν τους άφησε να προστατεύσουν αυτούς όπως πρέπει. Είναι βέβαια πολιτικό πρόβλημα. Όταν δεν έχει κανείς να τραφεί πρέπει να μπόρεσει να επωφεληθεί και χρειάζεται μια κάποια προστασία για την οικονομία. Αν τους προσφέρουμε αυτή την προστασία, ένα κάποιο είδος προστατευτισμού δηλαδή, τότε ουσιαστικά η επιτυχία τους περιμένει, είναι φαύλος κύκλος. Χρειάζεται να δούμε, να δούμε και οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να μιλήσουν για το μέα κούλπα τους. Η κυρία Σαργεντίντη και μετά Νόιζερ. Νομίζω ότι έχουμε κάπως καθυστερήσει στις εργασίες της. Γι' αυτό τρία λεπτά χρόνο μιλίας ο καθένας. Ευχαριστώ. Κατάλαβα το μήνυμά σας. Αυτές οι συζητήσεις για τον εμπέρο και την ανάπτυξη πρέπει να συναντούμε το ότι έχουμε κατά νου, ότι έχουμε και το άρθρο 208 της Συνθήκης ε, της Λισαβόνας, ε, ότι ε, ε, τουρκικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει ε, να εξαλείφουν στο αναπτυξικού στόχους που είναι η εξάλληψη της ανέχειας. Ε, όταν ε, μιλάμε για τον περίοδο, όταν μιλάμε για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, το εμπόριο αποτελεί ζωτικό τμήμα αυτής της δυνατότητας της εξάλληψης της στόχιας, αλλά και του αντιθέτου. Και αν δείτε τις ε, συζητήσεις για το εμπόριο, ε, λέγεται ότι το εμπόριο δεν είναι εξωτερικές υποθέσεις, όμως εμείς ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Σβέσον για την πολύ καλή έκθεση. Μία έκθεση η οποία μας δείχνει ε, πού μπορούμε να ωφελήσουμε όμως αυτό που με εντυπωσιάζει, που με εκπλήσει είναι ότι το Κοινοβούλιο πέρσι συζήτησε τη συνολική εμπορική στρατηγική με τον κύριο Ντεκούκτε και τώρα συζητούμε την εμπορική πολιτική για την ανάπτυξη. Αν το είχαμε κάνει σωστά την πρώτη φορά δεν θα χρειαζόταν να έχουμε εμπορική πολιτική για την ανάπτυξη. Θέλω να συγχαρώ και τον εαυτό μου, γιατί εσείς μόλις ψηφίσατε για τη δική μου έκθεση και είπατε ότι οι συμφωνίε οικονομικής εταιρική σχέσης με την Ανατολική Αφρική δεν θα έπρεπε να κυρωθούν από αυτό το κοινοβούλιο. Ξέρω ότι η Επιτροπή τα μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά, όμως εγώ υποστηρίζω, χαίρομαι πάρα πολύ που υποστηρίζετε τα όσα πιστεύω εγώ και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η συμφωνία οικονομικής εταιρική σχέσης δεν είναι καλή για αυτές τις χώρες της Ανατολικής Αφρικής. Τώρα, άκουσα την Κομισιόν που είπε ότι τα εμπόρια για το εμπόριο ε, δεν υπήρχαν για τις ε, ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο πρώτων υλών. Όμως εγώ θέλω να σας πω ότι έχουμε και πάρα πολλές ε, χώρες που εμπορεύονται τέτοιες ε, πρώτες ύλες ε, και να σας πω ότι άλλες χώρες δεν έχουν τα κίνητρα να αρχίσουν να μεταποιούν τα αγαθά για να δημιουργούν θέσεις εργασίας και για να ε, δημιουργήσουν καλύτερο εισόδημα για τους πολίτες, ε, γιατί είναι πάντοτε καλύτερο να εμπορεύεται κάποιος με ένα αγαθά από το να εξαγάγει πρώτες Και σε ό,τι αφορά τις, τα βιοκαύσιμα, είναι πρώτη γιατί η παραγωγή βιοκαυσίμων από τις οδιές ε, δεν γίνεται πολύ συχνά σε αναπτυγμένες χώρες. Σε ό,τι αφορά στα βιοκαύσιμα, ας είμαστε ειλικρινείς ναι, ναι, αν μου επιτρέψετε δύο ακόμη σχόλια και θα κλείσω. Λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς. στο βαθμό που συνεχίζουμε να διατηρούμε ε, το 5% των ε, βιοκαυσίμων ε, στην εδώ στην Ευρώπη, τελικά και εμείς συνεισφέρουμε στην εκρίζωση καλλιεργιών. Σας ζήτησα δύο σχόλια, Πρόεδρε, και να περάσω το τελευταίο μου σχόλιο, σας παρακαλώ. Έχετε ήδη καθυστερήσει 48 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, το ξέρω. Έχουμε και άλλες εργασίες. Καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι εγώ μη σκιώδη για τους πράσινου. Κύριος Νόισερ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σβένσον, τον εισηγητή. Ακούσαμε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων Μίτσελ Γκέρνς και Σαρτζεντίνη και ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι παρατηρήσεις ε, συμπληρωματικά. Ακούσαμε και όσα ελέγχθησαν από την Επιτροπή και από την Concord. Από την Επιτροπή και από την Concord θα ήθελα να είχα ακούσει πιο ξεκάθαρες διευκρινήσεις. Πολλά από αυτά τα οποία ε, είπαν και η Επιτροπή και η Concord ε, δεν ήταν επαρκή. Θα έπρεπε να γίνεται πιο συγκεκριμένα η συζήτηση, διότι τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την αναπτυξιακή μας πολιτική. Ε, άκουσα νομίζω από τον κύριο Γκέρενς ότι ε, δεν πρέπει να έχουμε ε, μόνο τα θέματα του Επιτρόπου για το εμπόριο, αλλά και τα θέματα ανάπτυξης. Λοιπόν, θα πρέπει και ο Επίτροπος Πίμπαλς να συμμετάσχει. Στις διαπραγματεύσεις και Ευρωπαϊκής Ένωσης είδα ότι δεν είναι πάντοτε ισότιμε οι διαπραγματεύσεις και όταν μιλάμε για ε, οικονομική εταιρική σχέση πρέπει να είναι ισότιμες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική εμπορίου και ανάπτυξης και θα πρέπει να συμμετέχουμε με, με ίσους όρους με τους εταίρους μας. Πιστεύω ότι ε, εδώ υπάρχουν πολλές προκλήσεις τις οποίες ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε την δυνατότητά μας για εμπόριο και θα πρέπει να δούμε όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ποσότητα. Να υπάρχουν δηλαδή κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορούμε να κρίνουμε αν ε, η καταπολέμηση της φτώχειας είναι κάτι το οποίο θα επιτύχουμε με την ενίσχυση του εμπορίου. Δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος δείκτης ε, που το προσδιορίζει αυτό. Άλλο ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι η μικροχρηματοδότηση, οι μικροπιστώσεις και ο ρόλος των γυναικών. Δεν το έχουμε τονίσει αρκετά αυτό και στις εταιρικές, οικονομικές εταιρικές σχέσεις και στις γενικευμένες ε, προτιμήσεις ε, θα πρέπει περισσότερο να εστιάσουμε σε αυτά τα θέματα και να συμπληρώσουμε την, τις παρεμβάσεις μας. Δεν έχω πολύ χρόνο και δεν μπορώ να επεκταθώ σε άλλες παρατηρήσεις. Ένα σημείο που θεωρώ σημαντικό είναι, ότι, είναι το εξής. Η Επιτροπή μίλησε και για τους φορολογικούς παραδείσους και είπε ότι έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια αρκετά δυναμικά. Εδώ θα πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπαθίες μας και εμείς ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Σβένσον. Έχετε το λόγο κύριε Σβένσον, αλλά να είστε σύντομος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και για όλες τις παρεμβάσεις ε, των συναδέλφων ε, και όλων όσων έλαβαν το λόγο. Από την Επιτροπή Ίντα θα ε, ξανασυζητηθεί το θέμα. Αυτό ήθελα να σας υπενθυμίσω και πολλά από τα σημεία τα οποία σήμερα αναφέρθηκαν θα συμπεριληφθούν και στο δεύτερο τμήμα που θα ακολουθήσει. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία έχουν ήδη επιτευχθεί, αλλά νομίζω ότι δεν είναι λάθος να επαναλαμβάνουμε κάποια πολύ σωστά θέματα. Η ιδέα δηλαδή του ότι πρέπει να έχουμε ισότιμη μεταχείριση των εταίρων μας και ότι θα πρέπει ε, να καταπολεμούμε τις, τους φορολογικούς ε, παραδείσους. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα και είναι και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία πρέπει να τονίσουμε και οι εξορυκτικές βιομηχανίες είναι ένα σημαντικό τομέα που πρέπει να τονιστεί. Όλα όσα ακούσαμε ήταν ε, σημαντικά και πρέπει να επαναλάβω ότι πολλά από αυτά τα οποία ακούσαμε ήδη υπάρχουν στην έκθεση. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι το εμπόριο δεν θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τις πλέον φτωχές χώρες. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι. Μιας και ο χρόνος μας πιέζει, θα συντομεύσω την παρέμβασή μου. Η βοήθεια για το εμπόριο είναι πολύ σημαντικό και για την Κίνα. Είναι κάτι που το χρησιμοποιούν οι Κινέζοι για να υποστηρίξουν τις επενδύσεις τους μάλλον παρά την ανάπτυξη. Τα σημειώνω λοιπόν όλα όσα ελέγχθησαν και ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Σβένσον και περνάμε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Ε, financier pluriannuel concernant le financement de la coopération de l'Union européenne en faveur... Εδώ τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ, την οικονομική συνεργασία και η χρηματοδότηση δεν εντάσσεται στα πλαίσια αυτή του προϋπολογισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γι' αυτό ακριβώς κρατιέται κάπως σε απόσταση από τις διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα το 2020. Γι' αυτό το λόγο συντάξαμε έκθεση πρωτοβουλίας και ο εισηγητής για το 11ο ΦΕΔ είναι ο κ. Πατρίς Τυρολιέν έχει το λόγο αμέσως για να μας εξηγήσει πώς έχουν τα πράγματα. Κυρία Πρόεδρο, σε ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Τρεις μήνες μετά από την υιοθέτηση της δικής μας τη θέσης ε, για τις διαπραγματεύσεις ε, για αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να δούμε και το μελλοντικό ΦΕΔ. Είναι το κύριο εξωτερικό μέσο βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε όμως δυστυχώς να πραγματευτούμε οτιδήποτε εδώ. Γιατί το εργαλείο αυτό, όπως θα το γνωρίζετε και πριν από λίγο είπατε, δεν είναι στα πλαίσια, δεν εγγράφεται στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα θα γίνει αυτό. Ελπίζω όμως ότι από κοινού θα συντάξουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο και θα το υποστηρίξουν οι περισσότεροι για να ακουστεί αυτή η φωνή από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η πρώτη μας συζήτηση γίνεται μετά από αυτή την ημερομηνία γιατί οι διαπραγματεύσεις για αυτό το πλαίσιο των πολιτές και με, ε, που θα συμμετάσχει και το ΦΕΤ δεν είχαν καταλήξει μάλλον αλλά σχετικά με το 11ο ΦΕΤ τα ποσά, τα εμπρικοδότησή του και η πρόσφατη προ πρόταση του πρόεδρου Βαμουμπή ήταν εντελώς απογοητευτική γιατί θέλει κατά 11% να μειωθεί το ποσό αυτό που πρότεινε η Επιτροπή. Και αν δούμε λεπτομερέστερα τις σημερινές προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος, η πολιτική ανάπτυξη υποφέρει περισσότερο από τις περικοπές του προπολογισμού. Πικρή η διαπίστωση τώρα που έτσι κι αλλιώς τα χρήματα αυτά δεν ήταν ποτέ αρκετά και από τους Ευρωπαίους πολίτες ε, τα τρία της βοήθειας έρχεται η βοήθεια στοχούς. Ε, να πούμε στα πλαίσια του, του επόμενου ΦΕΔ πρώτα απ' όλα να σημειώσουμε ότι θα είναι μετά τη συμφωνία Κότονου μια κάποια στιγμή που αναδιαρθρώνει σε βάθος ε, τη πολιτική της Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 10ο ΦΕΔ, ε, αλλά στο 2015 δεν θα υπάρχουν συγκεκριμένοι σαφείς ορισμοί σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της ανάπτυξης. Ε, ε δεν θα επαναλάβω εδώ τα όσα λέω στο έγγραφό μου το εργασίας, αλλά θα αρκεστώ σε αυτά που μου φαίνεται σημαντικά για την εργασία μας, για την το πώς θα μπει στον προπολογισμό του ΦΕΔ. Αυτό είναι το θαλάσσιο τέρας και χρειάζεται, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να μπει στα πλαίσια του προπολογισμού από το 2020. Αυτή η σημερινή λιτότητα όμως θα πρέπει να μας σωθήσει στην σοφία για να παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο το πολιετές. Δεύτερο σημείο τώρα με την εφαρμογή για τη διαφοροποίηση στα πλαίσια του ΦΕΔ. Ξεκινώντας δεν ήμουν και τόσο αισιόδοξο πάνω σε αυτό το θέμα αλλά μου επιβεβαίωσε ο Επίτροπος Πίμπαλ ότι η εφαρμογή στο 11ο φέντα αυτή της αρχής δεν θα έχει σαν συνέπεια τη μείωση του εθνικού προπολογισμού για τι χώρες ΑΚΕ, μέσες και ενώτερε. και πεπισμένο είμαι ότι με τη βοήθεια θα μπορούσαμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε αυτές τις χώρες για να προωθήσουμε, να αναπτύξουμε ε, διάφορα μέτρα κατά τις ε, φτώχειες για περισσότερη σιγουριά κλπ. Φορολογικά το ένα το άλλο. Γι' αυτό ακριβώς διατηρούνται, το διατηρηθούν οι εθνικές, ε, εθνικοί πόροι. Είναι πολύ σημαντικό σε οποιοδήποτε στο επίπεδο και για τον ιδιωτικό τομέα την στήριξη και για το πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά για τα προγράμματα αλλαγή. Χαίρομαι για την αρχική εργασία που έχει γίνει, όπως το αναφέρει και η έκθεση του κ. Γκέρενς. Ο νέος μηχανισμός αυτός κανονικά σαν στόχο κύριο θα πρέπει να έχει οι πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Υποστηρίζοντας τον ιδιωτικό τομέα σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί βοήθεια στον τοπικό ιδιωτικό τομέα και με αυτή την ε, συνδυασμένη προσπάθεια, με αυτό το μηχανισμό το πρόσφατο, καλούμε λοιπόν ε, την ε, Επιτροπή να κάνει μια μελέτη συνεπειών για να δούμε πόσο ο μηχανισμός αυτός θα βοηθήσει για να μειωθεί η φτώχεια, πώς θα βοηθεί το περιβάλλον, το οικονομικό κλπ. Και η συγκέντρωση των θεμάτων προτείνει Επιτροπή προς την καλή σωστή διάθεση πηγαίνει, αλλά στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ ίσως υπάρξει μια ερμηνεία ότι είναι ακριβώς ε, το συμφέρον μόνο και μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια γι' αυτό, ανάλογα με κάθε χώρα στην χάραξη μιας στρατηγικής, θα πρέπει να είμαστε υπέρ του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες και τους εταίρους μας και να λάβουμε υπόψη μας τις προτεραιότητές τους. Αυτή η συγκέντρωση των θεμάτων επίσης, κάτι που θα πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε, είναι ότι οι πόροι στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες δεν έφταναν έτσι κι αλλιώς ε, σύμφωνα με τις γνώμες για το 10ο ΦΕΝΤ ακριβώς. Για το OMD θα πρέπει να γίνουν πράγματα και χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Τροπή και στις χώρες ΣΑΚΕΑ και στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να δούμε το 20% του ΦΕΔ να πάει στην υγεία και την παιδεία όπως έγινε με το προηγούμενο πρόγραμμα. Επίσης ε, για τα υπερπόντια διαμερίσματα θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό και το ενίο πρόγραμμα θα πρέπει να δείξει τις νέες προτάσεις ε, για αποφάσεις που θα πάνε υπέρ αυτών των ε, περιοχών, το ΙΝΤΕΑΟ όπως το λέμε, όπως προτάθηκαν τον Ιούλιο που μας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καθόρισαν τους στόχους, ε, τους ε, περιοχών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο που είναι απαραίτητο για τις υπερπόντιες περιοχές με παρόμοιο επίπεδο ακριβώ από τις χώρες εκεί που είναι κάτι όμως απορχαιωμένο. Θα πρέπει να έχουμε τη φόληση να οικοδομήσουμε μια εταιρική σχέση που να βοηθήσει να αηφόρα ανάπτυξη των περιοχών αυτών, διαμερισμάτων αυτών, πάνω στον ανταγωνισμό και να συμφιλειωθούμε με τις αλλαγές του κλίματος και μια περιφερική συνεργασία ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ανυπομονώ να ακούσω τα σχόλιά σας και να μπορέσουμε με κάθε πολιτική ομάδα να συνεργαστούμε στενά και δεν ξεχνάω και την Επιτροπή με την οποία είχα καρποφόρες συναντήσεις και συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα ο κ. Γκέρεντς έχει το λόγο για δύο λεπτά. Γιατί σε πέντε λεπτά θα πρέπει να μα έλθει η Κύπρια Υπουργός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Στρούλιον ναι, χαίρεται που ακούει ακριβώς ε, όλα αυτά από τους συναδέλφους και να του πω ξεκινώντα ε, ότι δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μέσα από την πολλαπλή αυτή γλώσσα εδώ. Νομίζω όμως ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είχαμε αναλογή το 2005 για το 0,7% την ε, βοήθεια στην ανάπτυξη και δεν το κάναμε. Και μας λένε ότι θα μπει το ΦΕΔ στον προϋπολογισμό, θα ενταχθεί και τα κράτη-μέλη λένε ε, το κάνουν σαν να το είναι για αυτούς βέβαια αλλά όχι για τους υπόλοιπους και για την πρικοδότηση εδώ στο DCI και για την πρικοδότηση στα πλαίσια του ΦΕΔ για σαν είναι ένα σύνολο και μια υποχρέωση την αλλάζουν με πρικοδότηση σημαντική με το 2015 αλλά η υποχρέωση αυτή αλλάζει. Είναι μια μεταβλητή προσαρμογή στα προβλήματα τα σημερινά του προπολογισμού. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο που σημαίνει ότι αυτή η αλλαγή ε, σημαίνει και προδοσία για αυτή τη συνένεση του 2005. Προδοσία είναι, έτσι το αποκαλώ. Στην Επιτροπή Προπολογισμού πήγα και διαμαρτυρήθηκα για αυτή την κατάσταση και οπωσδήποτε θα συνεχίσω και με άλλους ε, θα πρέπει να, καταβάλ, να υποβάλω και μια τροπολογία ώστε τουλάχιστον από πλευρά μα ε, να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΦΕΔ και τι υπόλοιπες πολιτικέ ανάπτυξη, γιατί είναι κάτι το απαραδεκτό. Ενώ υπάρχει άρθρο που μας προσκαλεί να συντονίσουμε την όλη πολιτική, ουσιαστικά θα θυσιάσουμε ένα ακόμα μέρος της δημοκρατίας, δεν ασκούμε ιδιαίτερο έλεγχο προς το παρόν και σε αυτά τα λίγα που έχουμε ακόμα λόγο, τι θα κάνουμε, θα αφαιρέσουμε μέσα και εργαλεία και κατά την άποψή μου αποτελεί προδοσία αυτών των συμφωνιών και της όλης θεωρίας, αντίληψης πάνω στην οποία βασιζόμαστε για τη συνεργασία ο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Εντάξει, δεν ξέρω αν ε, θα το μοιραστούν το χρόνο για να λάβουν περισσότεροι τον λόγο και να εκφραστούν. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολο το έργο μου. Θα απαντήσω με διάφορα σημεία, γρήγορα-γρήγορα. Μου προσφέρετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την υποστήριξή του, όπως αυτή εμφανίζεται καθαρά στην έκθεση για τις προτάσεις της Επιτροπής. Συγγνώμη από τον συνάδελφό της Δακφός για τις υπερπόντες περιοχές που δεν είναι όμως εδώ σήμερα, ενώ θα το επιθυμούσε. Θα μιλήσω για μερικά σημεία όπως τα αντιμετώπισε και ο εισηγητής. για το πώς εντάσσεται στον προϋπολογισμό που είπαμε προηγουμένως συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή είπαμε το ενδέκατο να μείνει εκτός ε, προϋπολογισμού μέχρι το 2020 και να προετοιμαστούμε όμως για την ένταξή του τότε. και να μπορέσει να υπάρξει μια σύγκληση και όλα αυτά να γίνουν σε θελούσια βάση, να υπάρξει μια συνεργασία. Euh, λοιπόν, για τη σχετική διαφοροποίηση, ο ε, Επίτροπος Πλήμαξ μας επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν εθνικές ενισχύσεις ε, για τις χώρες ε, ΑΚΕ που το επιθυμούν και θα το λάβουμε υπόψη μας ε, για το πώς, ε, πού θα πάνε αυτοί οι πόροι ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν, ε, ανάλογα με τη διαχείριση, το ευάλωτο χαρακτήρα, τις νησιωτικές περιοχές, όλα αυτά και στα πλαίσια του 11 του ΦΕΝΤ, όπως ακριβώς προβλέπεται από το πλαίσιο του Κοτονού. Κάτι που θέλω να υπενθυμίσω Έστω και αν υπάρξουν ε, διαφορές με το νέα συνάντηση, δεν είναι κάτι το καινούριο. Στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης, ε, ε, του περισσότερου ευάλωτου και φτωχού, του υποστηρίζουμε πάντα όπως προβλέπονται από τη Συμφωνία του Κοτονού χωρί να λησμονήσουμε όμω και του υπόλοιπους. Άρα λοιπόν 2014-2020 στα πλαίσια τη συμφωνία. θα συνεχίζουμε να ε, ενισχύουμε με εθνικά περιφερειακά κονδύλια κλπ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα το συνδυασμό όλων αυτών των προσφορών δεν πρόκειται για ένα νέο εργαλείο, το χρησιμοποιούμε αρκετά χρόνια, αλλά είναι εργαλείο που θέλουμε να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, να διευρυνθεί και να καταλήξει σε μια χρησιμοποίηση να είναι μοχλός για τη χρηματοδότηση στο μέλλον. Προβλέπονται περαιτέρω μελέτες ε, για την ανάπτυξη του σχετικού εργαλείου. Για τη συγκέντρωση τώρα σε ενότητες. Θέλετε να διακόψω εδώ, ναι, για την κυρία Υπουργό. Ναι, διακόπτω λοιπόν. Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι, υποχρεώσεις έχουμε, είναι πολύτιμος ο χρόνο μας. Κύριε Μίτσελ, έχετε το λόγο για δύο το πολύ λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ πολύ για όλους έχετε δουλέψει γι' αυτό. Θέλω, παρουσία της Επιτροπής, να κάνω μια ερώτηση. Νομίζω ότι η συνοχή και ο συντονισμός ε, είναι δύο άλογα που βρίσκονται στον ίδιο στάβλο μεγαλύτερη συνοχή και μεγαλύτερο συντονισμό και τις αντίστοιχες εξοικονομήσεις που θα έχουμε και τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο αντίκτυπο που θα επιτύχουμε είναι κάτι το οποίο θα επιτύχουμε με μεγαλύτερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το έχουμε πει και στο παρελθόν γιατί μπορεί να προτείνει και η Επιτροπή, μπορεί να προτείνει και το Κοινοβούλιο αλλά χρειάζονται και οι Υπουργοί του Συμβουλίου θα μπορούσαν οι Υπουργοί του Συμβουλίου από μόνοι τους ναι, αν δεν τους ζητούν να λογοδοτήσουν τα εθνικά κοινοβούλια να μην επιτυγχάνουν πρόοδο αφού θα αγνοούν τις αντιδράσεις. Πρέπει λοιπόν και το Συμβούλιο να ε, συμμετάσχει στη μεγαλύτερη συνοχή και το μεγαλύτερο συντονισμό. Αυτό θα έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο με ό,τι αυτό σημαίνει για διάσωση ανθρώπινων ζώων, για βελτίωση της οικονομικής κατάστασης κλπ. Η Επιτροπή λοιπόν θα το λάβει αυτό υπόψη τη να βοηθήσει το Κοινοβούλιο, να μας βοηθήσει να συντονιστούμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, να έχουμε δύο φορές το χρόνο τέτοιες συναντήσεις όπου να μπορούμε να συζητάμε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τύριλεν. Δύο λεπτά για να ε, Κυρία Πρόεδρε, πολύ πολύ σύντομος. Πρόκειται για έγγραφο εργασίας. Άκουσα τις διάφορες τοποθετήσεις, παρατηρήσεις του κυρίου Γκέρενς τις παρατηρήσεις, ε, ιδιαίτερα ανάγλυφες. Θα τον συναντήσω και θα εξετάσουμε πώς αυτές οι παρατηρήσεις θα μπορέσουν να ενταχθούν στο τελικό κείμενο το οποίο θα συντάξω. τι είδα. Για διάφορα προβλήματα που εγώ έθιξα, για αυτή την διαφοροποίηση που έχουμε εξασφαλίσει σχεδόν, και οι περισσότερες, όλες οι χώρες θα υποφεληθούν από διάφορα κονδύλια, δεν θα τους στερηθεί η βοήθεια όπως σε μια πρώτη φάση πέθεται κανείς για τα υπόλοιπα δεν έχω κάποια παρατήρηση άλλη. Επαναλαμβάνω όμως, θα προσπαθήσω πάντα να συναντήσω, να συμφωνήσουμε, να μπορέσει να εξελιχθεί αυτό το έγγραφο εργασία και να δείξει, να συγκεράσει τις απόψεις όλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλήγω να σας πω ότι συνεχίζουμε την εργασία μας και από τον Ιανουάριο θα σας παρουσιάσουμε ένα έγγραφο με περισσότερες λεπτομέρειες και οριστικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Με δίτερ ευχαρίστηση στην Επιτροπή μας για δεύτερη φορά υποδέχομαι την κυρία Ερατό Κοζάκου Μαρκουλή, Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Στόχος της επίσκεψής σας είναι, εξ της κυρίας Καθρίν Αστονίπα, της εκπροσώπου Ένωσης για τις Εκδορικές Υποθέσεις, να μας πείτε για τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης αυτού του Συμβουλίου που είχε να κάνει με τη συνεργασία και την ανάπτυξη της 15ης Οκτωβρίου που μας πέρασε στο Λουξεμβούργο. Και σε αυτή τη συνάντηση οι υπουργοί συζήτησαν για την προετοιμασία μετά από το ΕΜΔ και μετά από τη συνάντηση του Συνήκωση και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφόρο ανάπτυξη, για αυτές τις μεταβαλλόμενες κοινωνίες και την προσέγγισή μας ε, για αυτά και χωρίς συζήτηση τρία συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα για την προσπάθεια της Ευρώπης με την κοινωνία πολιτών, δομέα των εξωτερικών σχέσεων, κοινωνική προστασία στην συνεργασία και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση αυτής της ανάπτυξης την ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε ένα από αυτά τα θέματα την Επιτροπή μας, κυρίως μετά το 2015 και το πώς με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε και θέλουμε εμείς την άνοιξη του 2013 να θεωτήσουμε την έκθεσή μας. Συντικά με την ανθεκτικότητα και σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, θα θέλετε όμως να πω ότι κάπως αμφιβάλλω κάποιο σκεπτικισμό, έστω και αν ε, αυτά που ανακοίνωσαν είπαν ότι σε αυτό εδώ ο στόχος ε, είναι να ε, υπάρξει μια αύξηση των κονδυλίων για το 2015 σε ποσό του ΑΕΠ, αλλά αυτούς τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι ό,τι παρατηρούμε πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση και εμείς με τα κράτη-μέλη διεξάγουμε αυτή τη σημαντική συζήτηση και γι' αυτό ακριβώς το στόχο θα θέλαμε να στείλουμε επιστολές ε, καλώντας τους Επιτροπούς Ανάπτυξης κάθε κράτους μέλους να επισκεφθεί την Επιτροπή μας. Κυρία Υπουργέ, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για τις εργασίες του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργός. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που παρευρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντα την ύπατη εκπρόσωπο τη Ένωση για Εξωτερικέ Υποθέσει και Πολιτική Ασφαλή, την κυρία Καθαρινάστον για να σα ενημερώσω για τα συμπεράσματα των συζητήσεων και για τη συνέχιση που θα δοθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα στι 15 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Όπως ε, πάντα ήταν ε, πολύ χρήσιμη η ευκαιρία για να έχουμε μια πολιτική που θα αφορά την χαράξη στρατηγικής ε, μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών Ανάπτυξη και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις υπηρεσίες της Κομισιόν για την εξαιρετική συνεργασία για την προετοιμασία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και κατά την ε, ίδια τη συνάντηση. Στη συνεδρίαση του Λουξεμβούργου τον Οκτώβριο είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία αποτίμηση της πρόοδου που έγινε σε κάποια νέα αλλά ιδιαίτερα κεντρικά ζητήματα πολιτικής όπως η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κοινωνίες μετάβασης και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην αδεκτικότητα. Το πιο σημαντικό είναι το εξής. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να εμπλακούμε σε μια συζήτηση για ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα αναπτυξιακά σήμερα, τη συζήτηση για το παγκόσμιο πλαίσιο μετά το 2015. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνά τα όρια της αναπτυξιακής πολιτικής και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Στην πραγματικότητα, σε ένα μεγάλο βαθμό, αφορά το τι είδους μέλλον θέλουμε και θα έπρεπε να εργαστούμε προς την επίτευξή του από κοινού. Επίσης, είναι ένα θέμα για το οποίο είμαι σίγουρη ότι και εγώ αλλά και εσείς θα επανέλθουμε πολλές φορές τα επόμενα έτη. Θα ήθελα να μάθω περισσότερο, περισσότερα για το ποιες είναι οι δικές σας, οι δικές σας απόψεις για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πριν ε, να αναφερθώ στο πρώτο θέμα της ε, ημερησίας διάταξης, ε, η ε, είπατε εκπρόσωπος, επίσης επιβεβαίωσε ότι οι μελλοντικέ ε, συναντήσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα προγραμματίζονταν ως ε, ξεχωριστές συναντήσεις που θα διαρκούσαν μισή ημέρα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένοι υπουργοί είχαν ήδη ζητήσει στο παρελθόν και η δέσμευση αυτή έγινε ευπρόσδεκτη από όλου στη συνεδρίαση. Να στραφώ τώρα στο κύριο θέμα της ημερησίας διάταξης, την διαδικασία κατόπιν των στόχων της χιλιετίας ε, και τη συνέχιση που θα δοθεί στην ε, διάσκεψη 2 συν 20. Η ύπατη εκπρόσωπος ε, τόνισε την προσωπική της δέσμευση για το θέμα και υπογράμμισε το πόσο Σημαντική είναι μία καθολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συζήτηση μετά το 2015 και για τη συνέχιση που θα δοθεί στη διάσκεψη Ρίο συν 20 που θα λάβει χώρα, που έλαβε χώρα μάλλον μας χωρίτε φέτος τον Ιούνιο. Συντονισμός ε, για τη συνέχιση μετά το Ρίο έγγραφο σχετικά με τη συνέχιση μετά το 20 κυκλοφόρησε και η κυρία Άστον αναφέρθηκε στην καλή συνεργασία που είχε με τους επιτρόπους Ποτότσινικ και Πίμπαλξ. Κατόπιν κάλεσε τον Επίτροπο Πίμπαλξ που είναι μέλος του πάνελ υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών να ενημερώσει ε, το σε, για την πρώτη συνάντηση του πάνελ που έλαβε το Σεπτέμβριο. Ο κύριος ε, Πίμπαλξ έκανε την ενημέρωση, αναφέρθηκε και στην ε, έκθεση που αναμένεται το Μάιο του 2013, τη συζήτηση που θα λάβει χώρα στη Γενική Συνέλευση των Εθνών το Μέο του 2013 και το έργο που συνεχίζεται στα πλαίσια του ΙΕ για τους βιώσιμους στόχους. Ως προς την ουσία, έδωσε έμφαση στο να διατηρήσουμε ε, την εστίασή μας στη μείωση της ανέχειας και στο να εργαστούμε προς επικαιροποιημένους στόχους της χιλιετίας που θα πρέπει να επικεντρώνονται σε ε, στην διακυβέρνηση, στην ισότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην αεφορία, στην καλή διαχείριση των φυσικών πόρων. Στη συζήτηση που επακολούθησε, σχεδόν και τα 27 κρατημέλη πήραν το λόγο δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν θα σα αναφέρω λεπτομερώς τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών, αλλά θα υπογραμμίσω κάποια κύρια ζητήματα που ανέκυψαν. Καταρχήν, οι Υπουργοί συμφώνησαν ευρέω με τις κύριε προτεραιότητες ε, που περιγράφονται στην ε, έκθεση του ΙΕ, δηλαδή να, οι νέοι στόχοι τη χιλιετία, να οικοδομηθούν γύρω από του τρει πυλώνε τη αηφόρου ανάπτυξη οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής και ειρήνη και ασφάλεια και διακυβέρνηση. Τυχές σχετικές με αυτά. Δηλαδή, να διατηρηθεί η εστίαση στη μείωση της ανέχειας, αλλά να διευρυνθεί η προσέγγιση και σε άλλα ζητήματα που επίσης είναι κρίσιμα για την ανθρώπινη ευημερία και την εφοροανάπτυξη. Δεύτερον, ενώ κάποιοι υπουργοί προτίμησαν ε, ένα απλό σύνολο ευνόητων στόχων. Κάποιοι ήθελαν μια πιο οριζόντια προσέγγιση που να αντικατοπτρίζει την αλληλεξάρτηση των διαφορών τομέων, το νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα κτλ. Και δημογραφία, ειρήνη, ασφάλεια, μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτον, Πολλοί υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για στενή συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας, των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα σε θέματα που αφορούν και την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση. Τέταρτον, πολλοί υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για καθολικούς στόχους που να μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες αλλά να είναι προσαρμοσμένοι σε περιφερειακό πλαίσιο και στην τοπική πραγματικότητα. Οι σχέσεις ε, δωρητών ε, δικαιούχων που στηρίζουν το σημερινό πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας θα πρέπει να αντικατασταθούν με κάτι πιο ισορροπημένο και πιο καθολικό. Τέλος, κάποιοι υπουργοί αναφέρθηκαν στο νέο πλαίσιο μετά το 2015 και είπαν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάποια ευάλωτα κράτη όπου υπάρχουν σειράξεις και αναφέρθηκαν σε ένα New Deal όπως ε, ανέφερε και το έγγραφο ε, του 2011 σχετικά με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Σε ό,τι αφορά τώρα στη διαδικασία και στην πορεία που θα ακολουθηθεί προς το μέλλον προς το 2015, οι Υπουργοί επίσης τόνισαν κάποια κύρια ζητήματα. Υπήρξε συνένεση υπέρ μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. κρατημέλη κράτη-μέλη ζήτησαν, είπα, ότι η και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πολλοί υπουργοί επίση τόνισαν την ανάγκη να αναπτυχθούν θέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε στενή συνεργασία με τους κύριους διεθνείς εταίρους, τις οργανώσεις και ομάδες κρατών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους στρατηγικούς εταίρους και στις χώρες BRIC, καθώς και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τη G77 και τις χώρες της υποσαχαρίας Αφρικής. Εδώ έχουμε διδάγματα από το Ρίο. Επίτροπος Πίμπαλξ και πολλοί υπουργοί επίσης πρότειναν να συμπεριληφθεί ε, το θέμα της διαδικασίας μετά το 2015 και στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου το 2013. Το δεύτερο κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεταβατικές κοινωνίες όπου η συζήτηση έλαβε χώρα βάσει μιας κοινή ανακοίνωση από την ύπατη εκπρόσωπο και τους επιτρόπους Πίμπαλξ και Φίλε. Στις αρχικές της παρατηρήσεις ε, η κυρία Άστον αναφέρθηκε στην πρόταση, στην κοινή ανακοίνωση και την έθεσε στο, κοινό, στο συνολικό πλαίσιο μιας ευρύτερης προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό ήταν να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των μέσων που διαθέτει να μπορεί να προωθήσει καλύτερα πολιτική ελευθερία, κυβερνήσει που θα λογοδοτούν, ε, αξιοπρεπής θέσης εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στις διαδικασίες ε, μετάβασης και σε κοινωνία σε μετάβαση. Ο Επίτροπος ε, Πίμπαλξ υπενθύμησε ότι η μείωση της ανέχεια παρέμενε κεντρικό ζήτημα στις διαδικασίες μετάβασης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο που χορηγεί τη βοήθειά της προκειμένου να διασφαλίσει πιο υφόρα αποτελέσματα. Οι Υπουργοί καλωσόρισαν ε, την ε, ε, κοινή ανακοίνωση κυρίως σε ό,τι αφορά τις εμπειρίες μετάβασης σε κοινωνίες μετάβασης. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις παρεμβάσεις του κάθε υπουργού, αλλά θα παρουσιάσω κάποια κύρια σημεία. Καταρχήν, οι υπουργοί τόνισαν ότι η εμπειρία και τα διδάγματα που κερδίθηκαν από την ίδια τη διαδικασία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην ε, διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ ε, της διαδικασίας μετάβασης. Ε, το European Transition Compendium, αυτή η επιτομή είναι μία πηγή πολύ χρήσιμη που πρέπει να χρησιμοποιείται πιο συστηματικά. Δεύτερον, καθώ όλε οι διαδικασίε μετάβαση ήταν διαφορετικέ, υπήρξε ανάγκη για προσέγγιση αναπερίπτωση βάση της κατάστασης και των αναγκών και των προτεραιοτήτων των χωρών εταίρων. Υπήρξαν επίσης προτάσεις ε, για να συμπληρωθεί η προσέγγιση more for more με μια προσέγγιση less for less στις χώρες εταίρους που δεν είχαν καλά αποτελέσματα στον τομέα της διακυβέρνησης. Τρίτον, οι υπουργοί τόνισαν το σημαντικό ρόλο της τεχνικής βοήθειας και της οικοδόμησης ικανοτήτων στις χώρες εταίρους, προγράμματα αδελφοποίησης και μέσα όπως το ΤΑΓΕΞ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρύτερα και αποτελεσματικότερα. Τέλος, υπήρξε γενική υποστήριξη για καλύτερο συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω κοινών αξιολογήσεων, κοινών αποστολών και κοινών προγραμμάτων. Η ύπατη εκπρόσωπος συνόψισε τη συζήτηση και πρότεινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να προετοιμαστούν βάσει τη συζήτηση που έγινε με του υπουργού. Τώρα αυτά τα συμπεράσματα είναι υπό Το τρίτο και κύριο σημείο τη ημερησία διάταξη αφορούσε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ανθεκτικότητα η συζήτηση έγινε βάσει μια ανακοίνωση τη Κομισιόν που είχε εκπονηθεί από κοινού από τους Επιτρόπου Πίμπαλξ και Γεωργίευα. Είπατε εκπρόσωπο Εισήγα εισήγαγε το θέμα αναφερόμενη στην επιστημιστική κρίση στο Σαχέλ και στο κέρας της Αφρικής που υπογράμμισε την ανάγκη για μακρινή μακροπρόθεσμη και συστηματική προσέγγιση για να δημιουργηθεί η ανθεκτικότητα. Τόνισε την ανάγκη για μια καθολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν βοηθούμε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα των ε, τοπικών και περιφερειακών δομών που αντιμετωπίζουν εσωτερικά ή εξωτερικά σοκ όπως φυσικές καταστροφές, ενόπλες σειράξεις, πολιτική αστάθεια, κλιματική αλλαγή και οικονομική κρίση. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερα εξοπλισμένη τώρα κατόπιν της δημιουργίας ε, της ε, Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Κρίση και των μέτρων ε, που λαμβάνει για την ανταλλαγή πληροφοριών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Η Επίτροπος Γεωργίευα κατόπιν παρουσίασε τις λεπτομερείς προτάσεις στην ανακοίνωση, τονίζοντας συγκεκριμένα την αποτελεσματικότητα του κόστους ε, της βελτίωσης της ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους. Τρία διαφορετικά σημεία ε, ήταν ε, πολύ σημαντικά. Καταρχήν, το να προκαταλαμβάνουμε την κρίση. Δεύτερον, μέτρα έκτακτης ανάγκης. Και τρίτον, ενίσχυση της ικανότητας απάντησης οι πρωτοβουλίε ΣΕΡ και ΑΖΙΡ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραδείγματα ότι αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Οι υπουργοί και η σημερινή αλλά και η μελλοντική Προεδρία του Συμβουλίου καλωσόρισαν την ανακοίνωση και υποστήριξαν πλήρω την πρωτοβουλία για την αρθεκτικότητα. Άλλοι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη να ενδυναμωθεί ο δεσμό μεταξύ τη ανθρωπιστική βοηθεία και τη αναπτυξιακή συνεργασία και να διατηρηθεί ευελιξία στο στάδιο του προγραμματισμού. Θέματα που έχουν να κάνουν με την επιστημιστική ασφάλεια, την αξιολόγηση κινδύνου και την αποτελεσματικότητα του κόστου των παρεμβάσεων και των πολιτικών τονίστηκαν από όλους τους υπουργούς. Είπατε εκπρόσωπος έκλεισε με μία αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη της Ομαλίας στο Μαγκαντήσιο που υπήρξε ανάγκη για μία καθολική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα ανθεκτικότητας, ασφάλειας και πολιτικής αστάθειας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστώ να προσπαθήσω να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Πούργο. Ο κύριος Κασμάρεκ έχει το λόγο. Πάνη Przewodnicząca, Szanowna Pani Minister. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να έχουμε αυτή τη συνάντηση μαζί σας. Αυτή η παράδοση των συναντήσεων κατά το τέλος της Προεδρίας είναι ιδιαίτερα θετική. Έχω μια ερώτηση και και ένα σχόλιο. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Ζολή στην αρχή, θέλω να συνεχίσω λέγοντας κάτι. Στα συμπεράσματα υπάρχει για άλλη μια φορά η επιβεβαίωση από τους υπουργούς ότι οι δεσμεύσει μα θα υλοποιηθούν και είναι η επιβεβαίωση από τη δήλωση και τη 19 η Ιουνίου φέτος. Και μου δίδεται η εντύπωση ότι από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο δεν έγιναν και πολλά που θα μπορούσαν να μας κάνουν να πλησιάσουμε στο στόχο αυτό. Χαίρομαι με το περιεχόμενο των συμπερασμάτων, αλλά ανησυχούμε αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Η επανεπιβεβαίωση των στόχων είναι πολύ σημαντική, είναι μια πολιτική δήλωση, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους. Γι' αυτό κάνω λοιπόν και την ερώτησή μου. Βλέπετε να υπάρχουν δυνατότητες να επιτύχουμε τους στόχους. Και άλλο ένα σχόλιο. Το Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση για τη συμφωνία μεταξύ Πρασίνου ε, Ακροτηρίου ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίου. Εγώ ε, επισκέφθηκα το Πράσινο Ακροτήριο όταν έφτασε ο πρόεδρος Μπαρόζο για να υπογράψει τη συμφωνία στο Πράσινο Ακροτήριο. Ήταν μεγάλο γεγονός για τη χώρα αυτή η επίσκεψη και αυτή η συμφωνία και συνέπεσε με την ε, πέμπτη επέτειο της υπογραφής της συμφωνίας με το Πράσινο Ακροτήριο. Μερικές φορές στην Ευρώπη δεν καταλαβαίνουμε πώς αντιλαμβάνονται οι εταίροι μας αυτές τις συμφωνίες. Και εγώ το έζησα ο ίδιος. Έζησα αυτό τον μεγάλο ενθουσιασμό και τον σεβασμό που τρέχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ε, συμφωνία αυτή και ευχαριστώ το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίαση που μας κάνατε για το, τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Υπουργών. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Μου φαίνεται ότι είναι κάπως ηρωνικό το ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπαίνουν σε μία ύφεση που αυξάνει τις ανισότητες ε, μεταξύ των πολιτών μας την ίδια στιγμή που οι Υπουργοί Ανάπτυξης κατανοούν πόσο σημαντικό είναι για την καταπολέμηση της φτώχειας να μειωθούν οι διαφορές με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, υπάρχει μια δόση ηρωνίας είναι κάτι το οποίο το βλέπουν έξω από την Ευρώπη, αλλά δεν το βλέπουμε μέσα στην Ευρώπη. Πώς ε, η κρίση δεν μας ε, βοηθά να κατανοήσουμε τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν της παρατήρησης αυτής, Θέλω να πω ότι συμφωνώ με τις βασικές αρχές που αναφέρατε. Ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, η φόρος ανάπτυξη. Αυτές είναι οι βασικές αρχές που βρίσκονται και πίσω από την πρόταση DCI που διαπραγματευόμαστε τώρα και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, συμφωνούν επί των αρχών ε, και θα συζητήσουμε για τη διατύπωση μεμονωμένων φράσεων. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Η ερώτησή μου είναι η εξής συμφωνούμε επί των γενικών αρχών, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Στη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης σχετίζεται με αυτό. Θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μεγάλη μείωση στον προϋπολογισμό για τις αναπτυξιακές πολιτικές και το DCI και το Ευρωπαϊκό ε, Αναπτυξιακό Ταμείο μπορεί να αποτελέσουν θύματα των περιορισμών που επιβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ποια είναι η θέση σας επ' αυτού και τι συζητήσεις γίνονται μεταξύ των Υπουργών για το θέμα αυτό. Αυτή την ερώτηση είχα. Ευχαριστώ πολύ. Α, και κάτι ακόμη να προσθέσω, ίσως είδατε ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει ένας πειρασμός να μειώσουν τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη στη χώρα μου, στην Ολλανδία. Έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός σχεδόν κατά 25%. Ε, πραγματικά δυσάρεστη κατάσταση. Ο κύριος Γκένετς έχει το λόγο τώρα δεν ξεφεύγουμε από την ε, διάθεση να μιλήσουμε για οικονομικά, όπως τα έκαναν και οι δύο προηγούμενοι, δεν θα διστάσω να μιλήσω για παρόμοιο θέμα, αν και με ενοχλεί κάπως. Η κυρία Υπουργό, που τόσο ευγενικά έρχεται εδώ για να μας εξηγήσει το τι έγινε, δεν αξίζει αυτά που θα, που θα προσάψω. Εντάξει, εσείς ε, εκφράζετε και την άποψη της ε, Λέδη Αστον και ήδη που αποτελεί πρώτο σε σχέση με αυτό που είναι πριν από δύο χρόνια γιατί η προηγούμενη προκάτοχό σας ε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παρόμοιο. Αλλά πρώτα απ' όλα για ορισμένες συμφωνίες Μιλήσατε ότι θα πρέπει κανείς να δείξει υπεύθυνη στάση για αυτή τη διαφοροποίηση και συμφωνούμε και εμείς οι περισσότεροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι, ότι θα πρέπει να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη, αλλά στα συμπεράσματα όταν τα βλέπω, τα διαβάζω εδώ για τις 15 Οκτωβρίου του 2015 στο 6 είναι αριστούργημα έτσι, συμβιλικής αντιμετώπισης που έχει σχέση με τη χρηματοδότηση της βοήθειας για την ανάπτυξη. Θα πρέπει να τη διπλοδιαβάσουμε. Το Συμβούλιο των Υπουργών ε, βλέπει με ανησυχία ότι η δημόσια βοήθεια μειώθηκε για την ανάπτυξη αλλά Είμαστε πάντα οι πρώτοι εταίροι σε παγκόσμιο επίπεδο, αληθεύει και μετά αναφέρεται κανείς για το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που τις 29 ε, Ιουνίου υπενθύμησαν ότι θέλουν ε, να φτάσουν να τηρήσουν την υπόσχεσή του 0,7% για το 2015. Αλλά εντελώς το αντίθετο γίνεται. Ορισμένα κράτη-μέλη και οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων πριν από 10 μέρε εκεί οπωσδήποτε θα το γνωρίζουν μετά από τις 29 Ιουνίου συνέβησαν διάφορα πράγματα σε χώρες, μειώθηκαν οι δαπάνες σε εθνικό επίπεδο και επίσης η πρικοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και επίσης ε, κάνουν δεκτή μία μείωση του DCI. Άρα λοιπόν παντού τα πάντα μειώνουν και μας λένε «Α, θα βοηθήσουμε πάντα αυτή τη βο... θα αυξήσουμε το επίπεδο για να φτάσουμε σε αυτό που προβλέπετε για το 2015». Αλλά θα χρησιμοποιήσουν τη διαέκφραση ε, μια έκφραση που χρησιμοποιούμε προηγουμένω. Μα δουλεύουν κανονικά. Τώρα, τι θα γίνει, μας λένε θα αυξήσουν ενώ μειώνουν. Και ακόμα πιο επιτιδευμένα μπορούν να τα εκφράσουν αυτά, αλλά δεν κρύβουν αυτό που συμβαίνει, ότι έχουμε βάλει όπισθεν. Είναι εντελώ απαράδεικτα για την, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Λέδη Άστον, την οποία εδώ εκπροσωπείτε νομίζω ότι συμμετέχει στις συνεδρίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ακριβώς. Θα πρέπει να τους πει που είναι εντελώς αντίθετη με τα όσα δήλωσαν ε, τον Ιούνιο του 2012. Έρχονται σε αντίφαση. Συνοχή είναι και αυτό, συνοχή της πολιτικής ε, σχετικά με τις ε, υποσχέσεις, με τις προηγούμενες δηλώσεις, με τη συνοχή, με τους στόχους, τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Εδώ θα πρέπει να ενισχύθει κάτι. Το έχει κάνει σίγουρα η Κιλέδη Άλστον, αλλά για να το δείξει καλύτερα θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή τη συνένεση στην ευρωπαϊκή της ανάπτυξης και αυτός το όλο πρόγραμμα για την ε, ανάπτυξη έχουμε προσκαλέσει και για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι είναι πίσω από εκείνη και ότι είναι εκείνη μπροστά, προπορεύεται για να υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια ό,τι έχει αποφασιστεί. Ελπίζω το Κοινοβούλιο, ελπίζω ότι δεν θα υποχωρήσουν ούτε ένα πόντο στα όσα έχουν συμφωνήσει γιατί εδώ στα επιχειρήματα, στο σημείο 6 της δήλωσης, ακριβώς ε, θα πρέπει να το επιθυμίσουμε. Αυτό που τους ζητάμε δεν είναι ούτε λιγότερο περισσότερο. Να σεβαστούν από τις 29 Ιουνίου υποστήριξαν στο Λουξεμβούργο και μετά από μερικές εβδομάδες τα πρόδωσαν αυτά. Όλα πάνε καλά μέχρι την προδοσία τι θα γίνει. Θα πρέπει να τη δούμε αυτή την προδοσία, να την ε, αγνοήσουμε, να μην ισχύσει. Έτσι για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Η κυρία Υπουργό έχει το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα των τριών ε, συναδέλφων. Ε, me... Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες δεν κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα και θα συγκληθεί άλλο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις αρχές Ιανουαρίου του 2013 από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Βαν Rompuy. Στι αρχέ λοιπόν του 2013 θα προσπαθήσει αυτό το, συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει σε κάποια συμφωνία για το πακέτο των ε, πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη αυτές τις συμβαστικές λύσεις, ε, ούτως ώστε να συζητηθούν τα διάφορα συμφέροντα που υπάρχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα μέσα να παράσχει αποτελέσματα στα διάφορα προγράμματα συμπεριλαμβανομένης και της αναπτυξιακής συνεργασίας. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι το θέμα της αναπτυξιακής συνεργασίας έχει πολύ ψηλή προτεραιότητα στις συζητήσεις μας. Οι συζητήσεις γίνονται στο πλαίσιο τριμερούς διαλόγου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε αυτές τις συζητήσεις. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων τον Ιανουάριο. Αλλά η αναπτυξιακή συνεργασία είναι σαφώς ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τους στόχους ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη δέσμευση του 0,5% μέχρι το 2015 και η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 53,5 το 2015 έχει μειωθεί στο 53,1 το 2011. Αυτή η μείωση ε, φέρνει το συνολικό επίπεδο ε, αναπτυξιακής, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας στο 0,42% του ΑΕΠ, ενώ το 2010 είχαμε 0,44% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση και την κρίση στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη θέση της ως μεγαλύτερος διεθνής δωρητής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας πάνω από το μισό της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα κρατών μελών. Μόνο τέσσερα κράτη-μέλη έχουν επιτύχει το στόχο. Πέντε κράτη-μέλη κρατούν τις δαπάνες ε, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας το 2011 πάνω από τους ε, μεσοπρόθεσμους στόχους του 2010 και 18 κράτη-μέλη δεν έχουν επιτύχει τους στόχους τους και τις δεσμεύσεις τους. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να επιτύχουμε μια προσεκτική ισορροπία στα πολιτικά μηνύματα τα οποία δίνουμε. Οι πολιτικές δεσμεύσεις ε, έχουν ε, μεγάλη σημασία και το γνωρίζουν αυτά τα κράτη-μέλη. Αλλά το αν θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας εξαρτάται και από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Η οικονομική κρίση σαφώς έχει επιπτώσεις πράγμα που αυξάνει την ανάγκη για περισσότερο αποτελεσματική βοήθεια, ούτω ώστε να έχουν μεγαλύτερη αξία τα δαπανόμενα χρήματα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, και η Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτά νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το δεύτερο κύκλο ερωτήσεων τώρα. Ο κύριος Κάσμαν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ενημέρωση. Αν μπορώ να απαντήσω κι εγώ εντάχει, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κύριος Γκέρανς και δεν έρχεται ως κάποιος α, μη σχετικός, ήταν αρμόδιος υπουργό για την ανάπτυξη και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και στο Συμβούλιο και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με τόσα μας παρουσιάσετε, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι το Ρίο συν 20 δεν ήταν η επιτυχία που παρουσίασαν κάποιοι, ιδίω ε, αν το δείτε ως προς τα δικαιώματα των γυναικών. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπήρξε μείωση στον τομέα αυτό. Περιστολή και για την ανάλυση μετά το 2015. Μπορούμε να αλλάξουμε τη φράση έτσι λοιπόν αντί να τελειώνει πάντοτε με το και ανθρώπινα δικαιώματα. Μήπως να ξεκινήσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί πιστεύω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προαπαιτούμενο για την επίτευξη της αηφόρου ανάπτυξης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίζουμε το άτομο. Και επίσης ε, τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ενισότητα και ως προς το εισόδημα Πάρα πολλοί φτωχοί άνθρωποι ζουν σε χώρες μεσαίου εισοδήματος και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε πιο άμεσα στην ισότητα μεταξύ των εθνών και να έχουμε στόχους και δείκτες που θα απαιτούν περισσότερη ισότητα. Και να έρθω τώρα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. Η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για μετά το 2015 είναι ακόμη τώρα πιο σημαντικό από σήμερα από ό,τι πριν. Έχουμε ε, ουσιαστικά μια συμφωνία που περιορίζει το πόση σημασία δίνει αυτό το κοινοβούλιο ακόμη και στη συμπερίληψη ρήτρα για τη μη εισαγωγή διακρίσεων Επίσης, ε, ε, δεν περιλαμβάνεται κάποιες ρήτρε σε σχέση με το γενετήσιο προσανατολισμό. Δεν θα ήταν αυτό ανησυχητικό αν δει κάποιος τι συμβαίνει σε κάποιες χώρες όπως η Ουγγάντα, το Καμερούν και η Αλγερία. Υποτίθεται ότι έχουμε ένα μηχανισμό για ένα διάλογο αμοιβαίο, αλλά αν η άλλη πλευρά γυρίσει και μα πει εμά δεν μα ανησυχεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει λοιπόν αμοιβαιότητα, τότε δεν γίνεται και διάλογο, Έτσι λοιπόν θα με ενδιαφέρει να ακούσω τι πιστεύετε εσεί σε σχέση με την επικύρωση στα, επόμενα, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη για τη Συμφωνία του Κοτονού και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε το θέμα του γενετήσου προσανατολισμού, ε, της θρησκείας, της νόσου, το κατάσταση του HIV, ε, την ε, ταυτότητα των φίλων και εδώ ε, αυτή τη βδομάδα κάποιοι εκπρόσωποι από χώρες της Αφρικής ε, πήραν ε, ουσιαστικά κάποια, πήραν μία θέση ε, και αναφέρθηκαν στο ότι εμποδίζονται τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν σε κάποιες πολιτικές διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα και πρέπει να το εξετάσουμε. Εγώ έτσι εκφράζω τις ανησυχίες μου εδώ. Φυσικά θα συνεργαστούμε στενά με την Βαρόνια Άστον και με τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Κομισιόν. Αλλά αν δούμε τη στρατηγική μετά το 2015, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί γιατί αποτύχαμε ε, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία. Έχει να κάνει με τα χρήματα, με τα κονδύλια. Είναι απαράδεκτο τα κράτη-μέλη όταν είναι φανταστικά τα πράγματα οικονομικά να λένε ναι, θα δώσω το 0,7% του ΑΕΧΠ και όταν είναι δύσκολα τα πράγματα δεν μπορούμε να το δώσουμε, να λένε τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είχαν ε, δεσμευτεί για ένα ποσοστό, όχι για ένα ποσό ε, χρημάτων. Εγώ πρέπει να ξέρω γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπάρχει μακροπρόθεσμη ή φόρος ανάπτυξη. Επίσης, για το κονβίλι 4, για το υπήρξε μία πρόταση μείωσης 10% και μετά είδαμε αύξηση από τον κύριο Βαρομπόη στο 11%. Αυτό είναι παράδεκτο εκτός ε, και αν ε, δεν ε, κάνουμε τίποτα παρά να λέμε δωρεά λόγια και τελικά να παρουσιάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ κύριος Μίτσελ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Εξωτερικών για την παρουσίαση που μας έκανε σήμερα. Και επανέρχομαι στο σημείο με το οποίο έκλεισε την παρουσίασή της. Όντως, δαπανούμε 96 δισεκατομμύρια για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αλλά νομίζω ότι για τα χρήματα που δαπανούμε, η αξία που αποκομίζουμε είναι περίπου 80 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αν είχαμε καλύτερο συντονισμό και καλύτερη συνοχή γιατί και η Επιτροπή ίδια έχει πει ότι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε 6 δισεκατομμύρια κατέτος ή να έχουμε αντίκτυπο επιπλέον δαπάνης 6 δισεκατομμύριων ε, κατέτος. Δεύτερον, αυτήν την εβδομάδα βλέπουμε τι συμβαίνει στι Φιλιππίνες. 350 άτομα νεκροί, 450 αγνοούμενοι και μπορεί να αυξηθούν αυτά τα στοιχεία δεν επενδύουμε όσο θα έπρεπε στην ε, αντιμετώπιση καταστροφών. Χαίρομαι για αυτά που είπατε για την ανθεκτικότητα και μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε ε, ανταπόκριση σε περιοχές καταστροφών. Η πρόληψη θα μπορούσε να είναι ένα μέσο. Αντί να τρέχουμε όταν έχουμε καταστροφές νεκρούς και αγνοωμένους και καταστροφή μεγάλων κοινοτήτων, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια μικροπράγματα παραδείγματο χάρη το να βάλουμε σε πιο υψηλό ε, υψόμετρο σχολεία και νοσοκομεία ή ακόμη και να μαθαίνουμε στους ανθρώπους να κολυμπάνε. Ε, αν δεν κάνουμε τέτοια απλά πράγματα προληπτικά, πώς θα έχουμε καλύτερη απόδοση για τα χρήματα που δίνουμε. Δεν έχει τη σωστή αξία το ποσό που δαπανάμε λόγω της έλλειψης συνοχής, έλλειψης προετοιμασίας. Καλύτερα να επενδύσουμε στην πρόληψη παρά την αντιμετώπιση των καταστροφών αφού λάβουν χώρα οι καταστροφές και οι καταστροφές θα συνεχίσουν να γίνονται πάντοτε. Τώρα, και για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και προς την ε, είπατε εκπρόσωπο την κυρία Άστον είναι σημαντικό να το πούμε αυτό γιατί αυτό θα δώσει αξία στα δικά μας ε, στα χρήματα που δαπανούμε. Μεγαλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα λοιπόν χρειάζεται και αυτό θα χρειαστεί και απόδοση μεγαλύτερου ρόλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια για να υπάρχει καλύτερη λογοδοσία. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Συνεκτικότητα, Καλύτερο συντονισμό, Θα ήθελα λοιπόν, Υπουργέ, να σα ζητήσω να το μεταφέρετε και στην ΥΠΑΤΗ ε, εκπρόσωπο στην κυρία και στο Συμβούλιο Υπουργών. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νόησε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα ε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω ε, που έρχεστε για δεύτερη φορά στην Επιτροπή μας. Ε, λάβατε μέρος και στην, ε, στο Συμβούλιο για θέματα ΑΚΕ και ε, είναι σημαντικό το ότι έχουμε αυτή τη σημαντική εταιρική σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Το Συμβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για το 0,7 ανέφερε ο κύριος Γκέρενς και ο κύριος Κάσμαν ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι το, τα όσα ήθελα να πω και εγώ. Όσον αφορά τους στόχους μετά το 2015 και το τι θα κάνουμε από εκεί πέρα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι περισσότερα θα επιτύχουμε με μια κοινή ευρωπαϊκή θέση. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ νομίζω ότι έχει εξαιρετικές δυνατότητες και για τα θέματα αυτά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να μπορέσει με μία φωνή να εκφραστεί, ούτω ώστε και στην αναπτυξιακή πολιτική στην Ευρώπη να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα, μια πολύ καλή ένδειξη και για τους στόχους της χιλιετίας και για τις προοπτικές μας για το μέλλον. Ένα δεύτερο τώρα θέμα ε, που δεν έχει άμεσα σχέση με τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αλλά έχει σχέση με τη συνεδρίαση με τις χώρες ΑΚΕ Θέλουμε καλύτερες ε, σχέσεις ε, με την Κούβα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα στο Σουρινάμ και θα ήθελα να ακούσω τη δική σας εκτίμηση. Πώς βλέπετε τις καλύτερες, τις βελτιωμένες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα που είναι μέλος των χωρών ΑΚΕ που δεν ανήκει όμως στην ε, Ισομερή Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πώς υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία. Και δίνω τώρα το λόγο, λέει η Πρόεδρος, στον κύριο Γκέρεν, τελευταίος παρεμβαίνων. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για την απάντηση που μου έδωσε ο υπουργό, την σέβομαι. Δεν είναι εναντίον της χώρας σας. Γνωρίζω τις δυσκολίες σας στη χώρα σας, σίγουρα. Αλλά μου δημιουργεί πρόβλημα η απάντησή σας. Μιλήσατε στο δημοσιομενικό πολιετές πλαίσιο και στα πλαίσια αυτού ακριβώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι στα πλαίσια αυτά του πολιτικού πλαισίου. Είναι ξεχωριστός προϋπολογισμός. Πάει για εκτέλεση με εντολή της Επιτροπής. Αλλά η στάση είναι σαν να ήταν μαζί. Και πάει στα κονδύλια του Ταμείου ανάπτυξη, σαν να ήταν ακριβώς ε, μέρος της όλης δέσμης για εξοικονόμηση κλπ. Και αυτό τώρα στα πλαίσια του τριμέρους διαλόγου εδώ δεν έχουμε τίποτα, κάνει μια ανάμειξη ούτε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ε, αλλά μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μα και να πούμε ότι αυτό είναι αντίθετο με τι υποχρεώσει που έχουν αληφθεί. Αλλά για τον προπολογισμό δεν μπορούμε να το κάνουμε επισήμως. Σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω. Είπατε ότι 11 χώρες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. 16 μπορούν, το κάνουν. Από τις 16 ορισμένες αμφιβάλλουν, διστάζουν ιδιαίτερα. Και τώρα η σειρά όλων αυτών των χωρών που διστάζουν για να αυξήσουν την πρικοδότηση. Ποιες είναι αυτές. Είναι οι χώρες που λένε ότι είναι καθαρή συνεισφόρη. Ε, Δηλαδή λένε ότι, ότι όταν και δύο λεπτά πληρώνουμε παραπάνω, α, χάνουμε, χάνουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν, δεν πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει, επιμένω, να επανέλθουμε στη συνένεση για την ανάπτυξη. Εάν δούμε τώρα ε, τα συμπεράσματα και δεν έχουν τηρήσει τις υποσχέσεις. Θα πρέπει να σεβαστούμε τη συνένεση που επετεύχθη γιατί όλοι οι θεσμικοί πυλώνες τα έχουν υποστηρίξει αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και από τη στιγμή που κάτι τέτοιο θα γίνει εγώ επιμένω ότι αποτελεί προδοσία η πράξη μας, απαράδεκτη προδοσία, συγχώρητη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη. Και ακόμα κάτι, διστάζουσες χώρες. Από αυτές Έχουμε και χώρες που δεν έδωσαν σχεδόν τίποτα όταν ήταν θετική η οικονομική συγκυρία. Τίποτα δεν προσφέρουν, ακόμα λιγότερο όταν έχουμε αρνητική οικονομική συγκυρία. Τίποτα λοιπόν, τίποτα αυτές οι χώρες ε, ουσιαστικά δεν σέβονται τις υποχρεώσεις, δεν το επιθυμούν. Έτσι, αυτή, αυτή είναι η πολιτική ερμηνεία και θα πρέπει να υψώσουμε τον τόνο και τη φωνή μας. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω στην Lady Άστον ότι θα μεταφέρει τα όσα εμείς εδώ φρονούμε, έτσι, και ουσιαστικά ε, δεν εμπιστευόμαστε πια σχετικά με την βοήθειά τους στην πολιτική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργό, έχετε το λόγο και πάλι για τις τελικές παρατηρήσεις σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσο μπορώ τις πολύ σημαντικέ ερωτήσεις και παρεμβάσεις και σχόλια που ακούστηκαν ε, από εσά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά, είναι κάτι πολύ σημαντικό, η ρεχοκοκαλιά των όσων κάνουμε στην και συνεργασία όπως και η διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Και αν ε, παραδείγματο χάρη δείτε τις εξελίξεις στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και η διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο επίκεντρο και πάντοτε θα πρέπει να αξιολογούμε την και με συνεργασία με πολλές χώρες λαμβάνοντας υπόψη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα διόρισε έναν ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο κύριος Λαμπρινίδης, ο οποίος είναι ο ειδικός εκπρόσωπος Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν ε, τις εξελίξεις στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους. Για όσο ερώτησε ο κύριος Μίτσελ, συμφωνώ απόλυτα ότι ο συντονισμός ε, και η συνοχή και το streamlining των δαπανών μας και των κονδυλίων μας στην ανάπτυξη και συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο, όλο ένα και περισσότερο, επιλέγουμε τον κοινό προγραμματισμό. Είναι πολύ σημαντικό καθήκον αυτό για να έχουμε μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ακολουθούμε μια νέα προσέγγιση, καλύτερος ε, συγχρονισμός και ευθυγράμμιση με τους εταίρους και τα κρατημέλη. Το 2001 είχαμε σημείο επιτυχία στην υπόθεση του Νοτιού Σουδάν. Και τώρα ξεκινάμε ένα κοινό προγραμματισμό σε πολλές χώρες εταίρους. Για φέτος κινούμαστε με την ε, Αιτή, το Λάος, το Μαλί, τη Ρουάντα, την Κάνα, την Αιθιοπία και επίσης διερευνούμε και άλλες δυνατότητες όπως η Βερμανία. Επομένως, ε, μέσω του κοινού προγραμματισμού τα χρήματα που θα δαπανίσουμε θα είναι ουσιαστικά πιο ευθυγραμμισμένα και θα υπάρχει καλύτερος συντονισμός και συνοχή. Αυτή είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε. Για να προσπαθήσουμε να δαπανίσουμε τα κονδύλια. με το δυνατότερο συνακτικό τρόπο για την Κούβα. Στο τελευταίο συμβουλίο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, οι Υπουργοί συζήτησαν ε, το θέμα αυτό και το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν ότι είπατε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, θα εργαστεί για διαπραγματευτικές οδηγίες για μια πιθανή νέα συμφωνία μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο Φυσικά, παραμένουμε με την κοινή θέση του Ινδέξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε ότι θα εργαστούμε για μια πιθανή νέα συμφωνία με την Κούβα. Προς στιγμή παραμένει η κοινή θέση. Και πατή εκπρόσωπος και οι υπηρεσία εξωτερική δράση θα εργαστούν για την κατάρτιση διαπραγματευτικών οδειών για μια πιθανή νέα συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στρατηγική μετά το στόχο ε, η ανακοίνωση Τη είπε τη εκπροσώπου είναι υπό και θα πρέπει να δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Υπήρξε και ένα ακόμη σχόλιο για τη μη εισαγωγή διακρίσεων ε, στο γενετήσιο προσανατολισμό. Όπως σωστά αναφέρθηκε, ήμουν και εγώ στο Σουρινάμ, στην κοινή συνεδρίαση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Χωρώνα και. Και φυσικά τέθηκε αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Όπως γνωρίζετε, υπήρξε μία πρόταση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού προκειμένου να μπει μια αναφορά και στο γενετήσιο προσανατολισμό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε αποδεκτό από τις χώρες ΑΚΕ. Ο συμβιβασμός που επετεύχθη ήταν ότι θα επικαιροποιηθεί η ρήτρα μη εισαγωγής διακρίσεων. Αλλά φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεδρίαση αυτή είχε την ευκαιρία να επαναλάβει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε μια διόρθωση. Η αναθεώρηση έχει συμφωνηθεί και τώρα περιμένουμε την ε, επικύρωση από κάποια κράτη-μέλη, από 12 κράτη-μέλη υπουργού και το Κοινοβούλιο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο διαπραγματευτής μας δέχτηκε ότι ε, δέχτηκε να υπάρχει γενετήσιο προνατολισμός, όμως οι χώρε ΑΚΕ δέχτηκαν ότι δεν συμπεριλαμβάνεται κάτι τέτοιο, που συμφωνήσαμε επί μιας διαφωνίας. Ναι, ναι, και εγώ αναφέρα αυτό. Προτείναμε τη συμπερίληψη του θέματος του γενετήσιου προσανατολισμού, αλλά Ξέρετε, στι διαπραγματεύσει αυτέ ε, συμμετέχουν δύο μέρη. Αν το ένα μέρο δεν ε, δέχεται τη ρητή αναφορά, τότε θα πρέπει να βρούμε ένα συμβασμό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, αποδυναμώνει τη δική της θέση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ε, κύριε Υπουργός, ε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και γιατί ήρθατε εδώ και γιατί μας δώσατε αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Σας εύχομαι καλό τέλος της Κυπριακής Προεδρίας και σε σας καλές γιορτές Χριστουγέννων. Τις αξίζετε πραγματικά μετά από τους μήνες δουλειάς. Λοιπόν, η επόμενη μας συνάντηση Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου από τις 3 το απόγευμα τις 6.30 και Τρίτη 18 από τις 9 έως τις 12.30 το Δεκέμβριο πάντα, έτσι. Παρόλο που έχουμε κοντά εκεί τις διακοπές των γιορτών, θα είναι παρόντες σίγουρα αρκετοί βουλευτές.